Okay, I think we had better start. What are... Ωραία. Μπορούμε να ξεκινήσουμε ίσως. Okay. I believe we are on agenda. Είμαστε στο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Κάτι μεταξύ 8 και 9, 8.30 ίσως. Uh, Right, this is agenda item 9. 9. Προς μια ουσιαστική οικονομική και νομισματική ένωση. Και θα δώσω το λόγο στην Μαριάν. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Έχουμε καιρό βέβαια να ανταλλάξουμε απόψεις όσον αφορά τις ε, τροπολογίες ε, πάνω σε μια ουσιαστική οικονομική και νομισματική ένωση. Νομίζω όμως ότι παρόλα αυτά καλό είναι να συζητήσουμε την ε, έκθεση πρωτοβουλίας που ζητήθηκε βάσει του άρθρου 220 της Εθήκης και να καταλήξουμε σε ένα νομοθετικό κείμενο, σε ένα ψήφισμα νομοθετικού περιεχομένου που να αναθέτει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ορισμένα πράγματα. Μετά τον Ιούνιο, τη διάσκεψη κορυφή του Ιουνίου. Ξεκίνησε λοιπόν ε, αυτή η πρόταση, το ζήτησαν ε, οι πρόεδροι, ζήτησαν δηλαδή για τον πρόεδρο να κάνουμε αυτή την έκθεση πρωτοβουλίας. Ο χρόνος δηλαδή που είχα στη διάθεσή μου ήταν πολύ λίγος. Ε, ξεκινήσαμε λοιπόν την προσπάθεια να σχολιάσουμε χωρίς όμως να είχαμε καιρό να ετοιμάσουμε αρκετές τροπολογίες. Πάντως, όπως και να έχει το πράγμα, καλό είναι να κρατήσουμε το δικό μας το χρονοδιάγραμμα, δηλαδή να ψηφίσουμε την επόμενη Δευτέρα, 15 Οκτωβρίου, και γιατί είναι τόσο σημαντικό αυτό. Γιατί την ίδια ακριβώς αυτή εβδομάδα υπάρχει διάσκεψη κορυφής του Συμβουλίου όπου θα συζητήσουν πάνω στο σημείο με αυτό του Φαν Και γι' αυτό πρέπει να είμαστε έτοιμοι κι εμείς και να δώσουμε περισσότερη σάρκα και οστά στην θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κατά τα άλλα δεν νομίζω ότι έχουμε πολλά να πούμε, είναι ότι μπορεί να κάνει δικιά μας η Επιτροπή. Και τέλος, όσον αφορά την Οικονομική και την ε, Νομισματική Ένωση, πρέπει να ξέρουμε ότι αυτό είναι και η καρδιά του έργου μας εδώ. Τώρα αγαπητοί συνάδελφοι, γνωρίζετε ότι εκ παραλίλου με την έκθεση αυτή, εκ τέλος πάντων ότι πέρα από τη δικιά μας τη δουλειά, δουλεύουν και οι πρόσωποι μας στη διάσκεψη των Προέδρων και ετοιμάζουν ένα έγγραφο το οποίο πρέπει να εγκριθεί από τους Προέδρους των ομάδων. Το θέμα είναι τι επιλογές θα κάνουμε για να ενισχύσουμε ο ένας τις θέσεις του άλλου. Να μην υπάρχουν επικαλύψεις. Πιστεύω πάντως ότι μπορούμε και ότι έτσι θα ενισχύσουμε τις θέσεις μας. Περιμένουμε ακόμα όμως και κάποια άλλα πράγματα την έκθεση της Επιτροπής Δεγματικών Υποθέσεων. Ε, βάσει της ενισχυμένης συνεργασίας συνεργαζόμαστε μαζί για μία έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Προπολογισμών. Και εκεί πρέπει να ψηφίσουμε ακόμα τις τροπολογίες που έχουν υποβληθεί. Συνεπώς, τα 15 Οκτωβρίου ψηφίζουμε και η έκθεση έτσι θα πάρει την τελική της μορφή. Τώρα έρχομαι στις τροπολογίες. 839. Νομίζω ότι έχουν εδώ πέρα οι συνάδελφοι εμπειρία με εκθέσεις στις οποίες υποβάλλονται τόσες πολλές τροπολογίες. Είναι πολύ δύσκολο να βρει κανείς ε, το νήμα μέσα από τόσες πολλές τροπολογίες. Πολλές ώρες περνάμε για να τις εξετάσουμε Αυτό που προσπάθησα εγώ να κάνω βάσει της εμπειρίας που έχω από άλλες φορές είναι βάσει όλων των τροπολογιών που μου έχουν φτάσει να διατυπώσω ε, για κάθε ομάδα συμβιβαστικές προτάσεις. Έχω κάνει το 65% του έργου αυτού και ελπίζω σήμερα το βράδυ, δεν σας υπόσχομαι 100% αλλά σήμερα το βράδυ αν μη τι άλλο ελπίζω να τελειώσω και με τα δύο τελευταία κομμάτια ώστε να μπορέσουν οι σκιώδεις να ενημερωθούν και αύριο μαζί τους να δω τι συμβιβασμούς μπορούμε να διατυπώσουμε. Αυτό είναι ο στόχος μου, αν μη τι άλλο. Και μετά βέβαια και θα σας πω πώς προτείνω εγώ να ψηφίσουμε, γιατί αλλιώς θα είναι πάρα πολύ δύσκολη η ψηφοφορία. Ελπίζω να επιτευχθεί σύντομα συμφωνία και να μπορέσουμε έτσι να καταλήξουμε. Τώρα με το πρώτο τμήμα, με τις αιτιολογικές αναφορές. Πρέπει να ξέρετε ότι έλαβε υπόψη με όλη τη δουλειά που έχει γίνει και εδώ αλλά και αλλού όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κανομισματική Ένωση και υπόψη του τι γίνεται σε άλλα πλαίσια, αλλά από την άλλη πλευρά δεν πρέπει να φορτώσουμε υπερβολικά το κείμενο και γι' αυτό να ξέρετε ότι έχω αφαιρέσει πολλά πράγματα. Δεύτερον, στις αγωγικές παρατηρήσεις. Εδώ υπάρχει η αιτία της κρίσης, η σημερινή κατάσταση, εξηγούνται όλα αυτά. 160 τροπολογίες πάνω σε αυτό το κομμάτι που προσπάθησα να επεξεργαστώ και να καταλήξω σε ένα πακέτο συμβιβαστικών προτάσεων. Υπάρχει και ένα τρίτο πακέτο που είναι η Τραπεζική Ένωση. Εδώ το έχουμε συζητήσει και εμείς αρκετά. Οι συνάδελφοι που θα θυμούνται το αρχικό σχέδιο θα θυμούνται ότι το είχαμε διαβρύνει, είχαμε βάλει και τον ενιαίο μηχανισμό εποπτείας, είχαμε βάλει τους μηχανισμούς ε, εγγύησεων η Τραπεζική Ένωση σίγουρα είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες του κειμένου του Φαν Ρομπάλ και γι' αυτό θέλω να συζητήσω εδώ στην Επιτροπή μας με τους συναδέλφους και να καταλήξω μετά. Ίσως δεν είναι πολύ έξυπνο να μπούμε σε λεπτομέρειες όσον αφορά την πρόταση, τις νομοθετικές προτάσεις. Προσπάθησα λοιπόν να αποδυναμώσω τουλάχιστον κάποια πράγματα να τα διατυπώσει ίσως διαφορετικά, ώστε με το έγγραφο αυτό να μην μπούμε σε διαπραγματεύσεις με άλλα θεσμικά όργανα για πράγματα για τα οποία βρισκόμαστε σε νομοθετικές διαδικασίες μέσω της συναπόφασης. Να το ξέρετε. Δεν θέλω δηλαδή να αποδυναμώσουμε τη θέση μας. Και να λέμε σε όλους να κοιτάξτε κάντε παραπάνω αυτό εκείνο. Όχι. Οι τρεις ε, πτυχές περιλαμβάνονται πάντως, αλλά αυτό το οποίο τώρα πρέπει να γίνει είναι η πρόταση για το μηχανισμό εγγύσεων καταθέσεων ή για τα σχήματα εξυγίανσης. Σε αυτά να δώσουμε το βάρος που πρέπει στην έκθεση αυτή. Δηλαδή το νομοθετικό έργο είναι αυτό που με ενδιαφέρει πιο πολύ και μπορούμε να πούμε αργότερα μπορούμε να κοιτάξουμε και εκείνο και το άλλο κτλ. Στη συνέχεια έχουμε την Δημοσιονομική και Οικονομική Ένωση. Αυτά είναι τα πιο δύσκολα κομμάτια για να τα διατυπώσω σε συμβαστικέ προτάσεις. Θα προσπαθήσω πάντως. Και πρέπει όλοι να αποφασίσουν κατά πόσο θέλουμε μια ισχυρή πλειοψηφία ε, πάνω σε κάτι το οποίο θα στείλουμε στο Συμβούλιο και μετά να δούμε πώς μπορούμε να επεξεργαστούμε παρετέρω το θέμα για την Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Μπορούμε δηλαδή με μια μεγάλη πλειοψηφία να το κάνουμε, αλλά μπορούμε να το κάνουμε και με μια μικρότερη πλειοψηφία, αλλά τότε το κείμενο που θα φύγει από το Κοινοβούλιο θα είναι κάπως λιγότερο ισχυρό. Πρέπει λοιπόν να συμφωνήσουμε πάνω σε πολλά θέματα και να καταλήξουμε σε συμβιβασμούς, τους οποίους σας λέω θα προσπαθήσω εγώ να τους ε, διατυπώσω, αλλά για την Δημοσιονομική και Οικονομική Ένωση είναι δύσκολο. Όλοι πρέπει να βάλουν νερό στο κρασί τους για να πετύχουμε κάτι. Υπάρχει μετά ένα άλλο πακέτο, πέμπτο ή έκτο, που είναι η δημοκρατική νομιμότητα και η λογοδοσία. Υπάρχουν πολλές νέες ιδέες που προστίθενται εδώ και μπορούμε όντως να τις προσθέσουμε και να φτιάξουμε έτσι ένα ενδιαφέρον ε, άρθρο βάσει του κυρίου Γαλτιέρη, ο οποίος ε, προτείνει κάποια πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Και βέβαια θα έχουμε και συμβιβασμούς σε αυτά τα οποία ζητάμε στην Επιτροπή. Αυτή είναι η κατάσταση πραγμάτων. Φυσικά δεν θέλετε να σας σχολιάσω τώρα 839 τροπολογίες. Θα συνεχίσω τη δουλειά μου σήμερα το βράδυ και ελπίζω αύριο με τους σκιώδες να μπορέσουμε να κάνουμε ένα μεγάλο βήμα προς τα μπρος για να ε, βοηθηθούμε στην ψηφοφορία που θα έχουμε την επόμενη εβδομάδα. Στόχος μας είναι μια ισχυρή πλειοψηφία, να εγκριθεί η έκθεση αυτή ε, με μια ισχυρή πλειοψηφία και έτσι να πάει στο Συμβούλιο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα ο κύριος Γκόγχο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω καταρχήν να συγχαρώ την εισηγήτρια η οποία έχει αντιμετωπίσει το το έγγραφο αυτό και τα θέματα συγχρόνως που άπτονται της Τραπεζικής Ένωσης και όλα αυτά μέσα σε ένα πάρα πολύ στενό χρονοδιάγραμμα. Πολύ προσεκτικά εξετάσαμε τις τροπολογίες συμβιβασμού που αφορούν την ε, Ένωση, την Τραπεζική και τη Δημοκρατία και περιμένουμε τα υπόλοιπα με αδημονία για τις τροπολογίες. Αυτά τα οποία περιλαμβάνονται είναι γενικά αποδεκτά. Αυτό που μας δημιουργεί προβλήματα είναι αυτά τα οποία ελείπουν. Υπάρχουν σημαντικές ε, ελλείψεις για την Τραπεζική Ένωση, για την ε, Ευρωπαϊκή Τράπεζα και για το Ταμείο Επίλυσης, το οποίο θεωρείται σαν μόνιμη λύση. Και επίσης το θέμα της, ε, του διαχωρισμού των δύο ταμείων. Έχετε προσθέσει και ορισμένα, έχετε προτείνει ορισμένε προσθήκε, οι οποίε δεν περιλαμβάνονται. Το, την άδεια για τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητα και την εποπτεία από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Για τα θέματα δημοκρατία τώρα. Υπάρχουν ορισμένα στοιχεία τα οποία είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικά. Παραδείγματο χάρη, ο σεβασμό τη μεθόδου, τη κοινοτική ή τη ενωσιακή καλύτερα και των ενωσιακών θεσμών αλλά περαιτέρω υπάρχουν κάποιες ελλείψεις σε σημαντικά σημεία. Σε σχέση με το αρχικό σχέδιο έκθεσης, δεν προβλέπεται η ψηφοφορία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πριν από το Εαρινό Συμβούλιο του, της επόμενης άνοιξης. Επίσης, δεν συμπεριλαμβάνονται ορισμένα στοιχεία για τον δημοκρατικό έλεγχο της Τρόικας και για την ενίσχυση της θέσης του Επιτρόπου, που είναι αρμόδιος για τα θέματα του ευρώ. Στους άλλους ε, πυλώνες, τον οικονομικό και τον πυλώνα του προϋπολογισμού, θα περιοριστώ να πω ότι αυτό το οποίο για μας είναι η προτεραιότητα είναι το να συμπεριληφθεί μια κοινωνική ρήτρα, μια κοινωνική συνθήκη στο πλαίσιο αυτό. Εδώ δεν μπορούμε να αρκεστούμε στα οικονομικά και νομισματικά θέματα. Προτείναμε την τροπολογία 814 για να υποστηρίξουμε την ιδέα και ελπίζω ότι αυτή η τροπολογία θα γίνει δεκτή. Η άλλη μας προτεραιότητα είναι οι επενδύσεις. Οι επενδύσεις είναι απαραίτητες για την ανάκαμψη και την επάνωδο Και αυτό είναι κάτι το οποίο το έχουμε τονίσει και συζητήσει με τους άλλους σκιοδησίγητες. Ευχαριστώ. Thank Η Σοφή, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και εγώ θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για τις προσπάθειες που έχει κάνει και το γεγονός ότι μελέτησε 850 τροπολογίες σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα είναι ένα Ηράκλειο έργο. Ε, επίσης, όπως και ο προηγούμενος ε, ομιλητής, θα ήθελα να αναφέρω ότι η συγγήτρια προτίμησε να βγάλει ορισμένα ουσιαστικά στοιχεία στο αρχικό κείμενο σε ό,τι αφορά την Τραπεζική Ένωση. Εγώ δεν μπορώ να κρίνω βέβαια ποιο θα είναι το τελικό αποτέλεσμα των συμβιβαστικών τροπολογιών, γιατί μας λείπουν ακόμα αρκετά στοιχεία για την Οικονομική και Δημοσιονομική Ένωση. Αυτό όμως το οποίο έχουμε ενώπιό μας δεν έχει κάτι το οποίο είναι επιλήψιμο για μένα, κάτι το οποίο εγώ μπορώ να έχω αντίθετη γνώμη. Νομίζω ότι για όλα αυτά τα οποία αναφέρονται υπάρχει γενική συνένεση, γιατί τελικά είναι πολύ λίγα από αυτά τα οποία ήταν στο αρχικό κείμενο και στις τροπολογίες. Εγώ όμως δεν βλέπω πώς μπορούμε να ψηφίσουμε 839 τροπολογίες επαρκώς αν πρέπει να ψηφίσουμε την επόμενη εβδομάδα. Δεν έχω πρόβλημα να ψηφίσω λοιπόν αυτό το οποίο έχει προτείνει η συγγήτρια, αλλά στερείται γενικά ψαχνού, δεν έχει πολύ περιεχόμενο. Είναι μια στρατηγική επιλογή το να αφήσουμε τα θέματα τα οποία είναι αφιλεγόμενα για άλλες εκθέσεις, αλλά μετά πρέπει να αναρωτηθούμε ποια είναι και η προσθέμενη αξία αυτής της έκθεσης. Εγώ νομίζω ότι είναι κρίμα και από κάποια άποψη οι συμβαστικές τροπολογίες υπολείπονται ακόμα περισσότερο από τις προηγούμενες θέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δεν ξέρω λοιπόν πώς πρέπει να κινηθούμε, γιατί δεν έχω, όπως σας είπα, προβλήματα. Πρέπει να την ξαναδιαβάσω την έκθεση και την πήραμε μονάχα σήμερα το πρωί. Αλλά σας λέω, δεν έχω αντίρρηση σε αυτά τα οποία λέγονται, αλλά δεν υπάρχουν και πολλά τα οποία για μένα θα αποτελούσαν ένα ουσιαστικό μήνυμα προς το Συμβούλιο. Θα προτιμούσα να έχουν συγκεντρωθεί οι τροπολογίες γύρω από ορισμένες πτυχές και να υπάρχει ένα πολιτικό μήνυμα στην έκθεση αυτή. Πιστεύω ότι αν μπορούμε να πάρουμε ορισμένες αποφάσεις ουσίες για κάποια θέματα, τότε κατά την άποψή μου θα προχωρήσουμε λίγο περισσότερο. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν προτείνουμε τίποτα. Μιλάμε για ένα ενιαίο εποπτικό φορέα για την Τραπεζική Ένωση. Αλλά δεν λέμε αν αυτό ο φορέας θα πρέπει να απαρτίζεται από την Κεντρική Τράπεζα ή από κάποιον άλλο. Είναι φανερό ότι στο βραχυπρόθεσμο διάστημα θα είναι η Κεντρική Τράπεζα που θα παίξει αυτό το ρόλο, αλλά ίσως μπορούμε να συζητήσουμε και άλλες επιλογές και άλλες μακροπρόθεσμε λύσει και θα πρέπει να έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και να εκφράσουμε γνώμη για τα θέματα αυτά. Ο Φιλίπ Μαριάν. Άκουσες τους δύο πρώτους ομιλητές. Όλοι σε ενθαρρύνουν να κάνεις κάτι ακόμα πιο πολύ. Το ίδιο θα κάνω κι εγώ. Συμφωνώ μαζί σου ότι πρέπει γρήγορα να καταλήξουμε ώστε το συμπέρασμα μας να ληφθεί υπόψη στην συνάντηση του Συμβουλίου αλλά από την άλλη μεριά πρέπει να υπάρχει και ουσία. Πρέπει να συμφωνήσουμε πάνω σε αυτό. Δεν πρέπει να δώσουμε την εικόνα ενός κοινοβουλίου το οποίο τελικά δεν σκέφτεται τίποτα. Ξεκινάω λοιπόν από την Τραπεζική Ένωση και σε στηρίζω εδώ. Δηλαδή για μένα η συζήτηση για την αρχιτεκτονική της ε, εποπτείας ε, θα γίνει και στις δύο εκθέσεις, και στην Τραπεζική Ένωση και στην άλλη εκθέση. Οπότε δεν θέλω να γίνει δύο φορές. Το κεφάλαιο αυτό δεν είμαι σίγουρος ότι υπάρχει χώρος για να διατυπώσουμε έντονα και τις απόψεις μας για το σύστημα εγγύσεων καταθέσεων και για την εξυγίανση που τελικά σημαίνει την αποκαινού θέση του χρέους. Οπότε για το τραπεζικό τμήμα πρέπει να μιλάμε για τα επόμενα βήματα. Το θέμα της εποπτείας για μένα θα εξεταστεί στα δύο νομοθετικά κείμενα. Οπότε εδώ συμφωνώ μαζί σου ότι λίγο ή καθόλου μπορούμε να μην συζητήσουμε γι' αυτό, να εξοικονομήσουμε τις δυνάμεις μας, ε, να μην υπάρχουν επικαλύψεις. Δεύτερον, συμφωνώ με τα σχόλια του Λίεμ για το AGS ακριβώς. Άλλη μια φορά θα έλεγα ότι η έκθεση των Υπουργών Εξωτερικών, ιδίω για αυτό το θέμα, δηλαδή για την ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης, ε, βεβαιώνει αυτό που λέμε εμείς. Δηλαδή θέλει να δώσει το ρόλο στους δύο συνομοθέτες, όχι μόνο στο Κοινοβούλιο, για την διατύπωση της ετήσιας επισκόπησης της ανάπτυξης. Οπότε δεν είναι δυνατόν το Κοινοβούλιο να μείνει πίσω σε σχέση με αυτά που λένε οι 10 Υπουργοί Εξωτερικών, αντίθετα. Πιο φιλόδοξο ακόμα πρέπει να είναι. Έπειτα για την Οικονομική Ένωση. Ακόμα και βάσει του δικού σου του προσανατολισμού, πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι παραπάνω. Εμεί εδώ και καιρό προτείνουμε να ενισχύσουμε την πειθαρχία για τη στρατηγική 2020, δηλαδή να είναι δεσμευτική και να είναι επίση όρος όπως και το Σύμφωνο σταθερότητα και ανάπτυξη Και το ίδιο για τον έλεγχο των εθνικών προγραμμάτων ε, όπως λέει το άρθρο 121 και το 133. Και η Σιλβή το λέει στην έκθεσή της, οπότε και εδώ να δούμε θέλουμε να υπάρχει τέτοια επικάλυψη με την έκθεση της Σιλβή Κουλάρα, αλλά ίσως θα μπορούσαμε να βάλουμε κάτι για την αποκαινουθέση του χρέους. Έπειτα υπάρχουν και οι ρήτρε πασαρέλα και υπάρχει και το δίχτυ ασφάλειας για τους ε, νέους σε μεγάλη δυσκολία. Τέλος, αλλά αυτή είναι και η ουσία για μένα, η ομάδα Βέστερβέλε. Ίσως όχι ο Ρομπάου, αλλά Βέστερβέλε. Δεν ε, σκέφτεται με αυτόν τον τρόπο. Εγώ νομίζω ότι όλοι ξέρουμε ότι έχουμε φτάσει στα όρια των όσων μπορούμε να κάνουμε. Ε, χωρίς αλλαγή στη συνθήκη. Και δεν καταφέρνουμε να αλλάξουμε ε, τα πράγματα με τα οπτίν ε, κλπ. κλπ. Κάποια στιγμή πρέπει να σκεφτούμε πέρα από τη συνθήκη. Δεν λέω όπως κάναμε με το Stability Bonds, αλλά να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και με τη συνθήκη αλλά και πέρα από τη συνθήκη. Γιατί κάποια μέρα θα πρέπει αυτή τη συνθήκη να την επανεξετάσουμε και θα μας το ζητήσουν οι πολίτες αυτό. Αν λοιπόν θέλουμε να εισακουστούμε και δεν θέλουμε να κάνουμε μια ωραία εκθεσούλα για την οποία όλοι θα μας χαϊδεύσουν, πρέπει να έχουμε περισσότερο θάρρος. Ξέρεις ε, Μαριάν ότι θα σε στηρίξουμε αν το κάνεις και πας πιο μακριά. Πρώτη φορά άκουσα γαλλόφωνο που να προφέρει το όνομα του Φάνο Ρομπά με τόσο σωστή προφορά. Συγχαρητήρια, Λίμ. Ήβο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς να πω ότι είναι λίγο δύσκολο να συζητήσει κανείς το θέμα αυτό όταν υπάρχουν 800 ε, τροπολογίες, δυστυχώς για την κυρία Τάισεν, ευτυχώς για μένα βέβαια. Είναι δύσκολο να προχωρήσει κανείς ε, με τέτοιο τρόπο, αλλά είμαι βέβαιος ότι θα τα καταφέρει με σωστό τρόπο. Όπως όλοι σχεδόν, και εγώ κατέθεσα μπόλικες σε εισαγωγικά τροπολογίες. Ξέρετε ότι συνολικά υπάρχουν άνω των 800 τροπολογιών. Τίθεται λοιπόν το θέμα τι είδους συζήτηση θα γίνει γύρω από την Πιστοτική Ένωση και τι θα πρέπει να προσθεθεί στην πρόταση η οποία είναι στη συγκεκριμένη φάση έτοιμη να κάνω πέντε προκαταρκτικές παρατηρήσεις. Θα τις παρουσιάσω ανάλογα με την προτεραιότητα ακριβώς την οποία δίδω εγώ. Το πρώτο, η πρώτη ομάδα τροπολογιών, η οποία θεωρείται ίσως και η πιο σημαντική, είναι η έννοια του υπολόγου δημοκρατικά της διαδικασίας αυτής. Αν συζητούσαμε εδώ και λίγες εβδομάδες το θέμα, δεν νομίζω ότι θα υπήρχε θέμα γύρω από τον δημοκρατικό έλεγχο. Γιατί όλοι εδώ είχαν δηλώσει επανειλημμένα ότι βλέπουν με σαν κάτι το πάρα πολύ σημαντικό τον δημοκρατικό έλεγχο της διαδικασίας. Θεωρούμε λοιπόν ότι είναι ένα κεντρικό σημείο της συζήτησης και γι' αυτό θεωρώ ότι θα αναζητήσουμε και θα βρούμε τη σωστή διατύπωση η οποία ανακαλύπτει αν όχι όλο τον κόσμο, τουλάχιστον τη μεγάλη πλειοψηφία. Η δεύτερη ομάδα τροπολογιών, η δεύτερη ενότητα αν θέλετε, αναφέρεται στο σεβασμό των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας. Δεν είμαι επίσης βέβαιος εδώ πόσο εύκολο είναι να καταλήξουμε σε συμβιβαστικές προτάσεις εδώ. Όμως, μια λειτουργική πιστοτική ένωση, τουλάχιστον για ένα τμήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να σέβεται τις αρχές αυτές. Και αυτό θα πρέπει να φανεί και στις ψηφοφορίες τις τελικές. Η τρίτη ομάδα τροπολογιών θα πρέπει να κρατήσουμε το δικαίωμα στα κράτη-μέλη να ελέγχουν τις ε, δημοσιονομικές τους πολιτικές. Εδώ και λίγες εβδομάδες όταν συζητήσαμε ουσιαστικά για πρώτη φορά την πρόταση της αρχιτεκτονικής για αυτή την συγκεκριμένη λύση. Από την Τσεχία, σαν παράδειγμα, ακούστηκαν φωνές και είπαμε ότι η Κεντρική Τράπεζα της Τσεχίας, η Εθνική, είναι υπεύθυνη σύμφωνα με το Σύνταγμα για τον έλεγχο ε, των πιστοτικών δραστηριοτήτων. Και το θέμα είναι ποιος θα έχει την τελευταία λέξη για τον έλεγχο της νομισματικής πολιτικής σε χώρες των οποίων το νόμισμα δεν είναι το ευρώ. Πρέπει να λυθεί το θέμα αυτό. Τώρα για την φορολογική ένωση. Έχουμε συμφωνήσει εμείς με τη μορφή του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου έτσι όπως έχει προταθεί αλλά να διευκρινιστεί εδώ ότι οι κρίσιμες αποφάσεις σε επίπεδο εθνικού προϋπολογισμού θα πρέπει να παραμείνουν στα χέρια του Εθνικού Κοινοβουλίου. Σε κάθε κοινοβούλιο, σε κάθε κράτος μέλος ο βασικός νόμος, ο σημαντικός, ο κρισιμότερος νόμος σε αιτήσια βάση είναι θα έλεγα ο προϋπολογισμός και αυτό θα πρέπει να παραμείνει αρμοδιότητα των εθνικών κοινοβουλίων, κοινοβούλια τα οποία είναι πιο κοντά στους εκλογείς τους από ότι ε, ε, εμείς. Αυτές είναι οι τέσσερις πέντε ίσως παρατηρήσεις Είμαι βέβαιος ότι θα προχωρήσουμε σωστά και θα μπορέσουμε να φέρουμε κοντά τις απόψεις μας και να πω ότι εκτιμώ ιδιαιτέρως την πρόταση της κυρίας Τάισεν μια προσπάθεια πολύ καλή σε ένα πολύ δύσκολο τομέα. Δεν ξέρω αν υπάρχουν άλλοι σκιώδεις εισηγητές ή εκπρόσωποι σκιωδών που θα ήθελαν το λόγο. Δεν υπάρχει εκπρόσωπος της Γκουε ούτε των φιλελευθέρων. Περνάω λοιπόν τώρα. Ο Ρομπέρτο έχει το λόγο. Ευχαριστώ λέει ο κ. Γουαλτιέρη. Σήμερα το πρωί η Επιτροπή ΑΦΚΟ ψήφισε την γνωμοδότησή της. Έχουμε λοιπόν ένα κείμενο για σας. Έχω παρουσιάσει μια πρόχειρη ερασιτεχνική λίγο θα έλεγα περιληπτική μορφή της νομοδότησης αυτής που μπορείτε να διαβάσετε ώσπου να έρθει στα χέρια σας το τελικό κείμενο που ψηφίστηκε επαναλαμβάνω το πρωί. Μπορώ να σας δώσω κάποια πρώτα στοιχεία χρήσιμα για την προσπάθεια τη δική σας, κάποια στοιχεία σημαντικά της, ε, του πρωινού κειμένου Επιβεβαιώνεται καταρχάς ο σκελετός της πρότασης ψηφίσματος και σχετικά με τη διάρκεια ισχύω των υπαρχουσών συνθήκων ή τις αλλαγές της συνθήκες και αναφέρομαι εδώ στην ανησυχία του κ. Λάμπερτ να πω ότι αυτό είναι θέμα το οποίο ανήκει στις αποκλειστικές αρμοδιότητες της ΑΦΚΟ και στην ΑΦΚΟ η συζήτηση γύρω από αυτό θα γίνει σε βάθος και γι' αυτό ακριβώς και η κυρία Τίσεν δεν έχει εμβαθύνει αν θέλετε. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας νομίζω μπορεί να διευθετήσει το θέμα με σωστό και ισόρροπο τρόπο. Δηλαδή μέσω όλων των μέτρων τα οποία μπορεί να ληφθούν με τις υπάρχουσες συνθήκες προχωράμε αναγνωρίζοντας όμως ότι η ολοκλήρωση μιας πραγματικής νομισματικής ένωσης περιλαμβάνει μια μεταρρύθμιση των συνθήκων. Και επαναλαμβάνουμε ότι το, Κοινοβούλιο εδώ θα ασκήσει το δικαίωμα πρωτοβουλίας του, το οποίο δεν μπορεί βέβαια να ασκηθεί μέσω μιας νομοθετικής πρωτοβουλίας του Κοινοβουλίου, αλλά μέσω των κατάλληλων μέσων, μέσα τα οποία πολιτικά να είναι θα έλεγα ισχυρά. Εμείς θεωρούμε ότι τα μέτρα με τις ισχύουσες συνθήκες είναι απαραίτητα για να δημιουργηθούν οι πολιτικές συνενέσεις που θα οδηγήσουν σε έφετο χρόνο στη μεταρρύθμιση της συνθήκης που πρέπει να περάσει από την ομοφωνία του Συμβουλίου. Πιστεύω λοιπόν ότι χωρίς να αλλάξουμε πορεία μπορούμε να προχωρήσουμε με τα μέσα που θέτει στη διάθεσή μας η οικονομική και πολιτική διακυβέρνηση γιατί έτσι μόνο θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μία μεταρρύθμιση των συνθήκων. Πρέπει να προχωρήσουμε λοιπόν σε δύο φάσεις και αυτό είναι απολύτως συμβατό με τα προγράμματα τα οποία προβλέπει η κυρία Τάισεν. Αυτά θα τα δείτε λοιπόν στην έκθεση ΑΦΚΟ αναλυτικά. Για τα υπόλοιπα, παραπέμποντας βέβαια στο τελικό γραπτό κείμενο φαίνεται ότι υπάρχουν ορισμένα θετικά θετικές διαπιστώσεις γύρω από τον δημοκρατικό έλεγχο και τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην, δημοσιονομική, στην συγγνώμη, Τραπεζική Ένωση. Ε, υπάρχει, τίθεται εδώ το θέμα και της ετήσιας έκθεσης για την ανάπτυξη των κατευθυντηρίων γραμμών και την πιθανότητα μιας διαδικασίας μέσω κατεχωρήσεως πράξεων επί τη βάση του 97 γύρω από το θέμα ειδικότερα της Φορολογικής Ένωσης. Η ΑΦΚΟ λοιπόν με την δική της προσπάθεια αποδεικνύει ότι είναι δυνατόν και με τις ισχύουσες συνθήκες να αυξήσουμε σημαντικότατα τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Νομισματικής Διακυβέρνησης και έτσι να καλύψουμε μία από τις βασικές θα έλεγα ελλείψεις της υπάρχουσας αρχιτεκτονικής. Το θέμα αυτό έχει ήδη προταθεί και από τους ΣΕΡΠΑ, τους λεγόμενους εκπροσώπους των κοινοβουλίων των κρατών μελών, μετά από την πολυμερή πρόταση και συζήτηση που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα, μετά από την πρόταση, την πρώτη πρόταση των τεσσάρων ΣΕΡΠΑ, που θα τύχουν οι προτάσεις τους νομίζω στήριξη της αρμόδιας επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχω άλλους δύο ομιλητές στον κατάλογο μου. Η Ελίζα Φερέρα και ο Βόλφ Κλίντς. Υπάρχει κάποιος άλλος. Ο Βούρχαρτ. είναι Κάποιος άλλος. Όλα αυτά τα χέρια εμφανιστικά τελευταία στιγμή. Η Ελίζα. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ θα ήθελα να συγχαρώ τη Μαριάν και να την ευχαριστήσω. Είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπίσει κανεί ένα τόσο πολύπλοκο και τόσο εκτενές θέμα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Δεν θέλω φυσικά να επαναλάβω αυτά που είπε ο Λίαμ εδώ προηγουμένω σε σχέση με τη θέση της δικής μου πολιτικής ομάδας. Θα ήθελα απλώ να υπογραμμίσω τρία ή τέσσερα σημεία. <clears throat> Σήμερα υπήρξε και η ψηφοφορία της η γνωμοδότηση της Επιτροπής Συνταγματικών Θεμάτων και της Επιτροπής Απασχόλησης. Είναι απαραίτητο λοιπόν να δούμε ποιες είναι οι απόψεις των άλλων γνωμοδοτικών επιτροπών σε σχέση με το θέμα αυτό. Σε σχέση τώρα με την ακολουθητέα στρατηγική, εγώ πιστεύω απόλυτα ότι η θέση μας θα πρέπει να είναι σαφής ώστε να δώσουμε στο Κοινοβούλιο μια επαρκή ορατότητα σε σχέση με το να μπορέσουμε να συμβάλλουμε, να καθορίσουμε την ε, κατεύθυνση που θα θέλουμε να ακολουθήσουμε σε μεσοπρόθεσμο επίπεδο και ποια είναι η στρατηγική που θα πρέπει να ακολουθήσουμε. <clears throat> Γιατί αυτό που είδα από την πλευρά της Μαριάν ήταν μια ιδιαίτερη επιφυλακτικότητα δεν ξέρω αν έχω κάνει λάθος στην αντίληψή μου. Πιστεύω ότι υπάρχουν θέσεις που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ψηφίσει τα τελευταία χρόνια και οι οποίες θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να παρουσιάσουμε τη θέση μας με σαφήνεια, με επικοδομητικό χαρακτήρα και με μια σαφή εικόνα για το ποια πρέπει να είναι σε μεσοπρόθεσμο επίπεδο η εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είχαμε πολλές εκθέσεις οποίες έχουμε ψηφίσει η έκθεση παραδείγματος χάρη της Περβάνς Μπερές για την κρίση, η έκθεση για την τραπεζική κρίση, τα θέματα για τον ε, φόρο Τόμπιν, για την ε, δημοσιονομική <clears throat> ένωση κτλ. Υπήρξαν πολλές εκθέσεις οι οποίες έχουν γίνει και για την θέση από κοινού του δημόσιου χρέους. Δεν πρέπει να έχουμε ε, ένα μείγμα ένα αμάλγαμα από ασυνάρτητες θέσεις, αλλά πιστεύω ότι έχουμε αρκετή δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε όλα αυτά τα στοιχεία που έχει ψηφίσει το Κοινοβούλιο για να φτάσουμε και σε ένα σενάριο το οποίο να είναι και πιο φιλόδοξο από αυτό το οποίο μπόρεσε να, φέρει σε, να εγκρίνει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το οποίο έχει επικυρωθεί και από τους τέσσερις προέδρους των βασικών θεσμικών οργάνων. Η έκθεση του Κοινοβουλίου λοιπόν πια δεν μπορεί να περιοριστεί μόνο σε μια επανάληψη των νομοθετικών κειμένων, θα πρέπει να τα συμπληρώσουμε με μια μεσοπρόθεσμη αντιμετώπιση η οποία θα μετατρέψει την Ευρωπαϊκή Ένωση σε κάτι το οποίο θα έχει ένα χαρακτήρα που θα την επιτρέψει να αντιμετωπίσει αυτές τις προκλήσεις. Υπάρχουν αυτοί οι οποίοι λένε ότι πρέπει να προχωρήσουμε σε αλλαγή των συνθήκων. Δεν πρέπει να ανοίξουμε το κουτί της Πανδώρας σε σχέση με την αλλαγή των συνθήκων. Θα πρέπει προηγουμένως να τονίσουμε την απόψή μας και να φυσικά να επιφυλαχθούμε σε μια <clears throat> μελλοντική μεταρρύθμιση των συνθήκων στην κάλυψη των κενών και των ελλείψεων που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν στις τωρινές συνθήκες. Αλλά πριν φτάσουμε εκεί πρέπει να συζητήσουμε πρώτα για το όραμα που έχουμε για την Ευρώπη σε μεσοπρόθεσμο επίπεδο. Θα ήθελα λοιπόν να παροτρύνω τη Μαριά να έχει μια πιο φιλόδοξη αντιμετώπιση σε αυτή την έκθεση η οποία είναι θεμελιώδης χαρακτήρα και η οποία ανταμοκρίνεται σε πράγματα τα οποία έχουμε ήδη ζητήσει εμείς. Μια μακροπρόθεσμη εικόνα της Ευρώπης και τέλος θέλω να υπογραμμίσω τη σημασία του να υπάρξει και ένας πέμπτος πυλώνας ο οποίος να περιλαμβάνει και το σεβασμό των κοινωνικών δικαιωμάτων των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό πρέπει να είναι ένα μόνιμο στοιχείο στα βασικά κείμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να υπάρξει λοιπόν ο πέμπτος πυλώνας, ο οποίος περιλαμβάνει και τα κοινωνικά θέματα, αλλά γενικά το μήνυμά μου είναι, Μαριάν, ας είμαστε πιο φιλόδοξοι και να χρησιμοποιήσουμε όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία έχουμε στο προστάσιο όμως ως ψηφίσματα του Κοινοβουλίου για να έχουμε όχι μια ουδέτερη στάση, αλλά μια στάση η οποία να είναι πολύ πιο φιλόδοξη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Βολφ Κλίνς. Η συνάδελφός μας η Μαριάν είχε ένα δύσκολο εγχείρημα να φέρει σε πέρας να δημιουργήσει μια ηλιοτυπία κατά κάποιο τρόπο για την αυριανή Ευρώπη. Αυτό είναι ήδη από μόνο το αρκετά δύσκολο και θα είναι ακόμα πιο δύσκολο δεδομένου ότι οι τμήματα αυτού του τομέα που αντιμετωπίζει η Μαριαντή Τάισεν έχουν ήδη αντιμετωπιστεί σε προηγούμενες νομοθετικές εκθέσεις, όχι μονάχα σαν εκθέσεις πρωτοβουλίας αλλά και νομοθετικές και πολλά από αυτά τα στοιχεία έπρεπε να τα επεξεργαστεί κάτω από μια τεράστια πίεση χρόνου. Εγώ δεν ξέρω τι συμβαστικέ ε, τροπολογίε. Κάποιοι συνάδελφοι φαίνεται τα έχουν δει αυτά, αλλά εγώ δεν έχω δει καμία συμβαστική τροπολογία. Αν η Μαριάν όμω θέλει να αποφασίσει να περιορίσει την έκθεσή της και να περιοριστεί σε τομεί όπου δεν έχουμε εκφράσει κάποια γνώμη σε προηγούμενες ε, εκθέσεις, αυτό μου φαίνεται εξόχως λογικό. Έχουμε αντιμετωπίσει παραγωγικά το θέμα της διαχείρισης της κρίσης σε εκθέσεις όπως η εκθέση Hercmark. Εκεί όμως που δεν υπάρχει τίποτα το νομοθετικό από την πλευρά του Κοινοβουλίου είναι απαραίτητο να τονίσουμε τα σημεία τα οποία έχουν ειδικό βάρος κατά την απόψή μας και τα οποία πρέπει να τα λάβει υπόψη του και το Συμβούλιο. Τώρα τι μπορεί να κάνει το Συμβούλιο στους επόμενους μήνες, παραδείγματος χάρη το καθεστώς του ενιαίου επόπτη, το SSM, αυτά θα σφραγίσουν για ένα μακροπρόθεσμο διάστημα το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εάν υπάρχει επιτυχία σε αυτά τα μέτρα, ίσως σε δύο-τρία χρόνια μπορούμε να προχωρήσουμε σε μια νέα συνέλευση η οποία θα αλλάξει και τις συνθήκες. Γι' αυτό να μου φαίνεται πάρα πολύ σημαντικό εμείς ως Κοινοβούλιο να δημιουργήσουμε ένα υπόβαθρο και να εξασφαλίσουμε ότι αυτά τα οποία είναι υπό επεξεργασία να μην δημιουργήσουν αρνητικά αποτελέσματα για την Ευρώπη. Να μπορέσουμε λοιπόν να ενισχύσουμε την ε, Ευρωζώνη αλλά να αποφύγουμε κάποια κάποιες διαλυτικές τάσεις ή τάσεις διέρεσης της Ευρώπης. Κάποιοι νομοματείς λένε ότι εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο, ότι στον νέο μηχανισμό μπορούν να μπαίνουν τα κράτη-μέλη μόνο όταν είναι μέλη της ζώνης του ευρώ και αν θέλουν να μπουν εθελοντικά, πάλι δεν θα έχουν τα ίδια δικαιώματα με τις άλλες χώρες. Βέβαια, ξέρετε ότι όταν ρωτήσουμε δύο μονομαθείς την άποψή τους, παίρνουμε τρεις απόψεις. Αλλά εδώ θέλω να σας αναφέρω αυτό το οποίο έχω ακούσει από ένα συνεργάτη του Γερμανικού Υπουργείου Οικονομικών. Εκεί λένε οι νομομαθείς ότι μπορούμε να έχουμε τη δυνατότητα του opt-in, δηλαδή της εισόδου της εθελοντικής ε, άλλων χωρών με τα ίδια ακριβώς δικαιώματα όπως οι χώρες που είναι μέλη της Ευρώπης. Αν λοιπόν υπάρχει αυτή η δυνατότητα πρέπει να τη χρησιμοποιήσουμε να αποφύγουμε τη διαίρεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλες οι χώρες τουλάχιστον οι οποίες έχουν δεσμευτεί εν καιρό να γίνουν μέλη της ζώνης του ευρώ θα πρέπει να συμπεριληφθούν μέσα σε αυτό το μηχανισμό με τη διαδικασία του opt αλλά με ίσα ακριβώς δικαιώματα με τις άλλες χώρες του, της ζώνης του ευρώ. Αυτό είναι το πρώτο μου σημείο. Δεύτερον, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα βρούμε μια λύση η οποία θα μπορεί να γίνει αποδεκτή και από τους πολίτες. Εμείς ερχόμαστε με νέες έννοιες, νέες προτάσεις, νέους κανόνες, νέες ρυθμίσεις. Μπορούμε να φανταστούμε πάρα πολλές λύσεις, αλλά ξεχνάμε ότι όλα αυτά τελικά θα πρέπει να τα εξηγήσουμε και στους πολίτες και να γίνουν αποδεκτά από τους πολίτες, αλλιώς κινδυνεύουμε να αυξήσουμε τον ευρωσκεπτικισμό στην Ευρώπη. και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας οδηγήσει να σκεφτούμε λίγο καλύτερα. Ο, οι πολίτες δεν υποστηρίζουν πολλές φορές αυτά τα μέτρα γιατί θεωρούν ότι δεν λαμβάνει υπόψη ο κανόνας της επικουρικότητος. Αν αναλάβει λοιπόν αυτό το έργο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ω επόπτη, αυτό μπορεί να τη δώσει αρμοδιότητα μόνο στον τομέα τον τραπεζικό. Οι άλλοι τομεί έχουν διαφορετικό χαρακτήρα. Έχουμε κάνει και στο παρελθόν συζητήσεις για την εποπτεία <coughs> και υπάρχει η εντύπωση ότι δεν είναι μονάχα μεγάλη η διασύνδεση των τραπεζών μεταξύ τους, αλλά και μεταξύ τραπεζών, πιστοτικών ιδρυμάτων, ασφαλιστικών εταιριών κτλ. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε λοιπόν ότι αυτή η ενιαία εποπτική δομή στην Ευρώπη θα έχει, ορισ δημιουργηθεί με ένα τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί η εποπτική της ε, αρμοδιότητα να καλύπτει όλους τους άλλους αυτούς πιστοτικούς και ασφαλιστικούς τομείς και να μην έχουμε κινδύνους οι οποίοι θα αναδυθούν από τους υπόλοιπους πιστοτικούς οργανισμούς αν περιοριστούμε στις τράπεζες. Γι' αυτό εγώ υποστηρίζω τη Μαριάν να εστιάσει την ε, προσοχή της μόνο στους τομείς όπου μπορεί να προσθέσει κάτι περισσότερο και θα πρέπει να δώσουμε προτάσεις οι οποίες θα παροτρύνουν το Συμβούλιο να δράσει, αλλά δεν πρέπει να επανέλθουμε σε αυτά τα οποία έχουμε ήδη συζητήσει και εκφράσει γνώμη για αυτά μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η Σύλβη. Πολύ σύντομα, Μαριάν, πολλά έχουν ήδη υποθεί. Έχω να κάνω δύο παρατηρήσεις. Πρώτα απ' όλα καταλαβαίνω την ανησυχία σας που θέλετε να είσαστε όσο γίνεται πιο φιλόδοξοι. Μερικές φορές πρέπει κανείς να διαλέγει, να διαλέγει προτεραιότητες και όχι να θέλει να τα καλύψει όλα, ακόμα και θέματα για τα οποία έχουμε λιγότερα να πούμε. Τώρα κάτι όμω που σκέφτομαι και δεν το έχω συμπεριλάβει στι τροπολογίε εξαιτία των τελευταίων εξελίξεων για την ε, μετάβαση από αυτό που γίνεται ε, χωρίς αλλαγή της συνθήκης με αυτό που μπορεί να γίνει με αλλαγή της συνθήκης θα μπορούσαμε να προτείνουμε πριν οποιαδήποτε επαναδιαπραγμάτευση της συνθήκης να σκεφτούμε το θέμα της επικύρωσης. Ψύχραμα χωρίς να σκεφτόμαστε μία συγκεκριμένη χώρα, αλλά πριν να ξέρουμε πού είναι τα προβλήματα, να συμφωνήσουμε με ποιο τρόπο θα γίνει η επικύρωση, έτσι ώστε κάθε χώρα να μπορεί δημοκρατικά να λέει ναι ή όχι, ανάλογα με το τι θέλει, αλλά σε κάποια χώρα αν το νο, το όχι θα είχε καταστρεπτικές συνέπειες και αν δεν έχουμε σκεφτεί από πριν πώς θα γίνει αυτό, καλό θα είναι και αν ίσως θα μπορούσες να το βάλεις κάπου στην έκθεση. Με διπλή πλειοψηφία για παράδειγμα, ίσως όχι παντού, σε κάποια κείμενα το έχουμε χρησιμοποιήσει και εν πάση περιπτώσει από τώρα μέχρι τη στιγμή που θα διαπραγματευτούμε για τη συνθήκη να έχουν συμβεί διάφορα τα οποία να έχουν διευκολύνει την πορεία. Για παράδειγμα υπάρχει ένα κογκρέσο τώρα από το οποίο φαίνεται ότι θα προκύψει δημοψήφισμα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αλλά εν πάση περιπτώσει χωρίς να λέω ότι έχω μια χώρα στο νου να υπάρχει η δυνατότητα επικύρωσης όσοι θέλουν να μπορούν να ε, μπουν στο πλοίο και να συνεχίσουν και όσοι δεν θέλουν όχι, εντελώς δημοκρατικά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την Μαριάν Τίσεν. Εγώ βλέπω ότι έχει κάνει μια τεράστια προσπάθεια για να μπορέσει να καλύψει αυτό το εκτενές πεδίο. Κατά τη δική μου άποψη, το έγγραφο εργασίας της ε, χαιρετίζει, είναι, είναι θετικό σε σχέση με την Τραπεζική Ένωση και την προοπτική της. Όλα αυτά όμως μπορούν να γίνουν πραγματικότητα όταν εδράζονται σε μια σταθερή βάση. Και πάντα κατά τη δική μου άποψη υπάρχει μια σειρά από νομοθετικά θέματα τα οποία είναι απαραίτητα για την ασφάλεια των καταθέσεων, για την ανάπτυξη χρηματοπιστωτικών θεσμών και για την κεφαλουχική επάρκεια. Όλα αυτά δεν έχουν ακόμα κλείσει και εφόσον δεν έχουν κλείσει όλα αυτά τα νομοθετήματα δεν υπάρχει ακόμα αυτή η σταθερή βάση την οποία χρειαζόμαστε. Ελπίζω λοιπόν ότι θα μπορέσουν να προχωρήσουν αυτά τα νομοθετήματα γιατί χρειαζόμαστε αυτή τη βάση για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε μια πραγματική οικονομική ένωση. Πριν χτίσουμε την σκεπή πρέπει να φτιάξουμε τα θεμέλια του σπιτιού. Η Σίλβια αναφέρθηκε στη διαδικασία κύρωσης. Η δική μου πεποίθηση είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι ιδιαίτερα ρεαλιστικό να προχωρήσουμε σε νέες αλλαγές των συνδικών γιατί θα πρέπει να κυρωθούν από πολλά κράτη-μέλη και μάλιστα κράτη-μέλη στα οποία η πιθανότητα να υπάρξει αποδοχή αυτών των αλλαγών στη συνθήκη δεν υπάρχει. Γι' αυτό θα το θεωρούσα πάρα πολύ θετικό αν η εισηγήτρια δώσει την έμφαση στα θέματα τα οποία είναι υπονομοθετική επεξεργασία αυτή τη στιγμή. Και συμφωνώ με αυτά που είπε ο Βολφ Κλίντς για τα κράτη τα οποία δεν είναι στη ζώνη του ευρώ, γιατί ο κίνδυνος ο πραγματικός είναι να προχωρήσουμε σε μια διάσπαση της ζώνης Τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να προχωρήσουμε λοιπόν με μεγάλη ευαισθησία και προσοχή στα θέματα αυτά, αλλιώ κινδυνεύουμε να πάμε στη Λάθο. κατεύθυνση. Ένα άλλο στοιχείο λεπτομεριακό το οποίο είναι για μένα πολύ ενδιαφέρον είναι το θέμα του κοινού ταμείου εξασφάλισης των καταθέσεων. Κατά την άποψή μου αυτό δεν συνάδει με αυτά τα οποία ψηφίσαμε τον Φεβρουάριο εφέτος όταν είχαμε για πρώτη φορά αντιμετωπίσει το θέμα αυτό Εν είναι μια διαδικασία η οποία είναι ακόμα εν και συμφωνώ με άλλους σκιώδεις εισηγητές ότι αυτή η εξασφάλιση, το Ταμείο Ασφάλισης των Καταθέσεων θα πρέπει να είναι το τέλος της διαδικασίας. Και το... η επίτευξη αυτού του θέματος φυσικά σημαίνει μια κοινή ευθύνη και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο συνάπτεται με το κίνδυνο του ηθικού κινδύνου που μπορεί να δημιουργηθεί. Τεχνικά βέβαια όλα αυτά τα οποία προτείνονται είναι πάρα πολύ ε, ενδιαφέροντα και φιλόδοξα για να μπορέσουμε να κλείσουμε αυτό το θέμα. Εύχομαι κάθε επιτυχία στην εισηγήθεια για να μπορέσει να ξεμπλέξει το κουβάρι των τροπολογιών και να μπορέσουμε να ψηφίσουμε μέσα στο χρονοδιάγραμμα αυτό και είμαι και εγώ ε, έτοιμος να συμβάλλω στη δημιουργία συμβαστικών τροπολογιών πριν από την τελική ψηφοφορία. Ωραία. Ο Όλε. Ευχαριστώ. Έχω εμπιστοσύνη στην εισηγήτρια. Κατάφερε να καταλήξει σε συμβιβαστικές προτάσεις σε σχέση με το CTB. Το πρώτο αφορά τον δημοκρατικό έλεγχο και το υπόλογο Όλα τα έγγραφα τα οποία έχουν παρουσιαστεί τα τελευταία ένα-δύο χρόνια έχουν θα έλεγα αναφορές της δημοκρατίας πάρα πολύ συνοπτικά. Και αυτό είναι κάτι το αρνητικό, ενώ έχει μεγάλη σημασία να διασφαλίσουμε τη δημοκρατική νομιμότητα αυτού που κάνουμε και ιδιαίτερα αυτών των ενεργειών που άλλοι αναλαμβάνουν να κάνουν. Πρέπει να υπάρξει αύξηση του, του δημοκρατικού ελέγχου, γιατί αλλιώς θα δημιουργηθούν περισσότερα προβλήματα από αυτά που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Ένα άλλο θέμα είναι αυτό το ανέφεραν ήδη πολλοί συνάδελφοι. Ξέρετε ότι εγώ είμαι υπέρ της, α, ε, α, ε, του να μπει η Σουηδία στην Ευρωζώνη, είμαι στη μειοψηφία αυτό τον καιρό και δυστυχώ το ποσοστό των φίλων του ευρώ δεν αυξάνεται. Παρ' όλα αυτά μια περαιτέρω διέρεση της Ευρώπης θα είναι μια καταστροφή. Και δεν θα ήθελα να δω τις συνέπειες μιας τέτοιας διαδικασίας. Δεν θα πρέπει να λέμε ότι εμείς παραμένουμε με ανοιχτές τις πόρτες, εμείς θα πρέπει να ακούσουμε προσεκτικά και να συλλέξουμε προτάσεις οι οποίες θα μπορούσαν εν πολλής να γίνουν δεκτές από τις χώρες εκτός Ευρωζώνης. Και περιλαμβάνω εδώ και το Ηνωμένο Βασίλειο. Μπορεί να, να θυμώνεται με κάποιες από τις παρατηρήσεις οι οποίες έρχονται από τη Μεγάλη Βρετανία, αλλά θα ήταν καταστροφή αν κάποιες χώρες μείνουν, εξής, μείνουν εκτός. Μην τους δίνετε λοιπόν την δυνατότητα να πούμε κοιτάξτε τι συμβαίνει στην Ήπειρο και θα πρέπει να φύγουμε. Αυτό θα είναι καταστροφή. Όχι μόνο για το Ηνωμένο Βασίλειο, όπως λέει και η Πρόεδρος, αλλά και για όλους εμάς στις υπόλοιπες χώρες. Εγώ αυτό που λέω Σιλβί είναι να είναι κανείς δεκτικός απέναντί τους. Εγώ έχω ακούσει ορισμένες παρατηρήσεις οι οποίες ε, δεν, ε, δεν είναι θετικές. Όταν κάποιος σου βάζει τις φωνές δεν πρέπει να το αναποδίδεις. Άλλα λέει βίβλος βέβαια, εν πάση περιπτώσει. Εγώ δεν έχω πάρει μέρος στη συζήτηση αυτή παλαιότερα, έχω καταθέσει ορισμένες τροπολογίες με τον Τόρβαλτσεν, αλλά νομίζω ότι πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό σημείο και είναι τμήμα της συζήτηση που κάνουμε και στη δική μου χώρα. Ας μην δώσουμε την ευκαιρία σε αυτούς που λένε ότι α, δεν μας θέλουν στην Ευρώπη, οπότε δεν πειράζει θα τα καταφέρνουμε μόνοι μας. Αυτό θα ισχύσει στη δική μου χώρα και σε άλλες χώρες γιατί δυστυχώς ακούγεται. Λοιπόν, όλοι να είστε καλοί και όλοι να αφήσετε τις πόρτες σας ανοιχτές. Λοιπόν, εκτός από την εισηγήτρια θα πάρει κάποιος άλλος το λόγο. Έκμαρκ. Θα ήθελα κι εγώ να υποστηρίξω πλήρως αυτά τα οποία λέει ο κύριος Σμιτ. Μερικές φορές απογοητεύεται που δεν τον στηρίζω, αλλά σήμερα πρέπει να το πω. Όταν θέλουμε να συζητήσουμε θέματα ευρωπαϊκής εποπτείας, πρέπει να είμαστε πολύ σοβαροί. Κανένας δεν είναι κατά μιας καλύτερης μορφής εποπτείας και θα πρέπει εμείς να καταλήξουμε με ένα πρόγραμμα το οποίο να μην είναι χειρότερο από το σημερινό. Η πολυδιάσπαση εκφύσεως θα εξασθενήσει την ευρωπαϊκή οικονομία. Θα εξασθενήσει την ζώνη ευρώ, θα εξασθενήσει και το ίδιο το σύστημα ελέγχου. Δεν μπορούμε να έχουμε δύο διαφορετικά συστήματα ελέγχων. Θα πρέπει καταρχάς λοιπόν να διασφαλίσουμε λοιπόν αυτά τα οποία ήδη έχουμε στη διάθεσή μας και να προσπαθήσουμε να συζητήσουμε πώς θα αναπτύξουμε περισσότερο την κατάσταση. Μερικές φορές υπάρχει ανταγωνισμός για την δημιουργία νέων μορφών ενώσεων, ένωση σταθερότητας, ένωση οικονομική, ένωση και ακόμα και τα συνδικάτα παίζουν με το λέξεις trade union και union γενικότερα στα αγγλικά. Λοιπόν, εγώ θα είμαι πιο ριζοσπάστης. Πρόεδρε, γιατί να μην επενδύσουμε σε αυτό το οποίο ονομάζω πάρα πολύ απλά Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πολιτική, είναι οικονομική, είναι φορολογική, είναι ένωση της αγοράς, είναι εμπορική ένωση γιατί φυσικά εμπορευόμεθα ημέν με τους δε. Λοιπόν, ζούμε δύσκολους καιρούς. Πρέπει η ένωση να παραμείνει ένωση. Η πολυδιάσπαση είναι το χειρότερο που μπορεί να γίνει. Πρέπει να υποστηρίξουμε αυτά τα οποία πρέπει να βελτιωθούν και να κρατήσουμε ενωμένη την Ένωση. Νομίζω ότι όλοι μας αυτό το θέμα θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε με σοβαρότητα, να σκεφτούμε τις ευρωπαϊκές μας ευθύνε. Δεν το ακούω συχνά αυτό τελευταία. Ακούω πάρα πολλές προτάσεις οι οποίες δημιουργούν περισσότερη διαίρεση και όχι ενότητα. Εγώ θα ήθελα να ακούσω όλο τον κόσμο ε, για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι για το Βορρά, για τον Νότο, για την Ανατολή, για τη Δύση. Λοιπόν, θα πρέπει να τονίσουμε ότι η ένωση που χρειαζόμαστε είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακούγεται ριζοσπαστικό, αλλά αυτή είναι η δουλειά μας. Πρέπει λοιπόν να υπογραμμίζω ότι και ο Όλε Σμιτ συμφωνεί πλήρως μαζί μου. Ευχαριστώ πολύ. Η Μάριαν είναι υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Διάφορα πράγματα ακούστηκαν εδώ στη συζήτηση. Αρκετές φορές μιλήσατε για την τροποποίηση της συνθήκης και ότι μισοπρόθεσμα θα πρέπει να σκεφτούμε τι ε, μπορούμε να κάνουμε πέρα από την υπάρχουσα συνθήκη. Το είπα και στην αρχή όμως τη συζήτηση ότι ασχολούμεθα με μια έκθεση πρωτοβουλίας με ψήφισμα βάσει του άρθρου 225. Δεν μπορούμε λοιπόν να βγούμε από αυτό το πλαίσιο. Για τελειώς μπερδευόμαστε. Μπορούμε βέβαια να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έρθει με νομοθετική πρόταση. Τι τροποποίησεις πρέπει να γίνουν κτλ. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε και το έχουμε χρησιμοποιήσει και άλλη φορά να το κάνουμε και τώρα. Και αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινεί, έτσι κι πρέπει να τηρούμε τους κανόνες. Γι' αυτό εγώ δεν ξεκίνησα με την ιδέα αυτή για το τι μπορούμε να κάνουμε στο μέλλον ε, έχοντα προτείνει τροποποίηση των συνθήκων. Γιατί δεν ήταν ε, αυτό το οποίο ανέλαβα. Τώρα, για να πάμε πιο πέρα. Πώς θα επικυρωθούν δεχόμενες τέτοιες τροποποίησεις στις συνθήκες, αυτό είναι θέμα και των Εθνικών Κοινοβουλίων. Ε. Περισσότερο είναι δικό τους θέμα παρά δικό μας. Πρόεδρε, άκουσα διάφορες ε, ιδέες που και μένα ε, μ' αρέσουν, αλλά που χρειάζεται τροποποίηση της συνθήκης. Δεν νομίζω όμως ότι τώρα πρέπει να ασχοληθούμε με αυτά. Αλλιώ θα πρέπει να γράψουμε ολόκληρο βιβλίο για το μέλλον και δεν θα γράψουμε κάτι συγκεκριμένο, μια συγκεκριμένη πρόταση όπως θέλουμε προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν υπάρχουν πάντως πολλέ τροπολογίε που αναφέρονται σε τροποποίηση των συνθήκων. Τώρα για το πόσο φιλόδοξοι είμαστε. Είπα ότι θα προσπαθήσω όντω να κάνω συμβαστικέ προτάσει ομαδικά, παίρνοντα ομαδικά διάφορε τροπολογίε. Δεν έχει πολύ νόημα να καταλήξουμε ένα, δύο, τρία. Καλύτερα θα είναι να συζητήσουμε λιγάκι, ελπίζοντας βέβαια πώς θα καταλήξουμε τελικά σε συμφωνία. Χωρίς βέβαια να λείπουν τα ουσιώδη από μέσα. Ναι, σε συνένεση, σε συμφωνία. Όντως, στην πολιτική οι συνενέσεις δεν είναι τόσο ελκυστικές. Παρ' όλα αυτά πρέπει να καταλήξουμε σε συμφωνίες. Μερικές φορές έτσι και συμφωνούμε, άλλες φορές όμως είμαστε διχασμένοι και άλλοτε πολύ διχασμένοι. Εδώ, βάσει της συνθήκης του άρθρου 225 και το δικό μας κανονισμό, δεν πρέπει να έχουμε μια απλή πλειοψηφία, πρέπει να έχουμε μια απόλυτη πλειοψηφία στην Ολομέλεια. Και αυτό το λαμβάνω υπόψη μου και γι' αυτό και προσπαθώ πράγματι να καταλήξω σε προτάσεις που θα βοηθήσουν την Οικονομική και Νομισματική Ένωση, αλλά από την άλλη μεριά με τις οποίες θα συμφωνήσουν οι συνάδελφοι και δεν θα μας διχάσουν ακόμα περισσότερο. Προσπαθώ να πετύχω κάτι πάνω στο οποίο να μπορούμε να πούμε ναι, οι περισσότεροι από εμά το στηρίζουμε και αυτό να στείλουμε σαν μήνυμα προς τα έξω, προς το Συμβούλιο. Πολλοί υπογράμμισαν πόσο μεγάλη σημασία έχει η δημοκρατική νομιμότητα. Φυσικά και είναι πολύ σημαντικό, το υπογραμμίζω και εγώ. Γι' αυτό και λαμβάνω υπόψη μου την έκθεση Βαλτιέρη που περιμένω πώς και πώς και θα τη χρησιμοποιήσουμε. Κατά τα άλλα, θα συνεχίσω. Σας είπα τι θα κάνω με τις τροπολογίες, έτσι κι αλλιώς, όποτε έχουμε πολλές τροπολογίες, αυτό κάνουμε εδώ στο Κοινοβούλιο. Προσπαθούμε να τις ε, συμπεριλάβουμε σε συμβαστικές προτάσεις. Αυτό θα κάνω κι εγώ και ελπίζω ότι θα βοηθήσει. Πάντως, να ξέρετε κυρία Πρόεδρε, ότι δεν πρόκειται όλοι οι συνάδελφοι να είναι ενθουσιασμένοι, γιατί καταλαβαίνετε ότι δεν είναι εύκολη δουλειά. Κάτι ακόμα. Άκουσα πάρα πολλά, τα οποία δεν τα βρίσκω όλα στις τροπολογίες. Δεν πρόκειται να γράψω νέα συνθήκη, όπως καταλαβαίνετε, ούτε να ξεκινήσω από την αρχή την ε, έκθεσή μου, αλλά βάσει τον όσο να άκουσα θα προσπαθήσω να τη βελτιώσω. Ελπίζω ότι θα καταλήξουμε σε ένα αρκετά δυνατό κείμενο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος. Το χρονοδιάγραμμα προς το παρόν προβλέπει την ψηφοφορία στις 15 Οκτωβρίου και να πάμε στην Ολομέλεια του Νοεμβρίου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε περίπου 10 λεπτά πριν από την ψηφοφορία. Προβλέπω την ψηφοφορία στις 4.30 και θα κάνουμε μια μικρή διακοπή μέχρι τις 4.30 ε, διαφημιστικό διάλειμμα. Okay, can you take your seat? Λοιπόν, καθίστε παρακαλώ. Right, thank you very much. Um, λοιπόν, ε, έχει ζητήσει το λόγο... Ποιος? Α, παρακαλώ. Συνήθως καθώς αλλού. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να σας δώσω ένα καλό νέο. Μήπως δεν το γνωρίζετε κάποιοι από εσάς. Από ό,τι φαίνεται, σχετικά με την εισαγωγή του φόρου ε, συναλλαγών. Είναι μια ιστορική σημασίας απόφαση η οποία επιβεβαιώνει τις προσπάθειες που έχει κάνει το σώμα όλα αυτά τα χρόνια. Καλώς, ευχαριστούμε. Τώρα θα ψηφίσουμε. Μαριάννα, είναι η έκθεσή σου, ε, το Κοινό Ευρωπαϊκό Δίκαιο Πολίσεων. Σωστά. Είμαστε έτοιμοι για την ψηφοφορία. Θέλετε να ελέγξουμε, έχετε τις κάρτες σας. Βάλτε δε στο μηχάνημα. Αν κάποιος δεν έχει την κάρτα του να σηκώσει το χέρι για να καταλάβω εγώ δεν έχω για παράδειγμα, λέει πρόεδρος, άλλος κανείς. 33 κάρτες, 26 πάτησαν ε, το κουμπί όμως. Ε, οι υπόλοιποι, για πατήστε και εσεί κάποιο κουμπί για να δούμε αν δουλεύουν οι κάρτες σας καλά. Από τους σοσιαλιστές ένας παραπάνω εμφανίζεται. Ένας σοσιαλιστής πρέπει να βγάλει την κάρτα του. Τα μηχανήματα μου το λένε. Δεν σας μετράω... Α, εντάξει, τα έβγαλε κάποιος. Ωραία ο Ρόμπερτ. Καλώς. Οπότε, αρχίζουμε. Τροπολογία ρυθμός 10. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 8. Με προφορική τροποποίηση, πρώτα την, τρο... την προφορική τροπολογία, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία τώρα με την ε, τροποποίηση υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 12. Υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 13. Υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 14. Υπέρ, Α, όχι, 14 καταπίπτει. Συγγνώμη. 15 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 16 έχει αποσυρθεί. Συμβιβαστική δέλτα, D υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 18 τώρα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 19 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική α. Ε υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 21 υπέρ. Κατά. Έχει αποσυρθεί. Δεν υπάρχει στο δικό μου το χαρτί, λέει πρόεδρος. 21 έχει αποσυρθεί, από ό,τι φαίνεται. 22 τότε. Προφορική τροποποίηση. Πρώτα που προτείνει η Για την 22. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 22 τροποποιημένη υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική Β. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 25 με προφορική τροποποίηση, πρώτη τροποφορική τροποποίηση υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 25 τροποποιημένη τώρα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 26 και 27 έχουν αποσυρθεί και τώρα τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική γάμα C υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και τώρα ψηφίζουμε το τροποποιημένο κείμενο ηλεκτρονικά παρακαλώ. Πέρασε η να προσθέσουμε και τη δικιά μου ψήφο, οπότε είναι 34 υπέρ, τέσσερις κατά και καμία αποχή. Ευχαριστώ Μαριάν. Συνεπώς, η έκθεση της Αρλίν για τον ε, κανονισμό όσον αφορά την κατάχρηση της αγοράς. Είσαστε έτοιμοι να ψηφίσουμε. Ωραία. Συμβιβαστική Α. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική Β. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική γάμα σι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική δέλτα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική ε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική Έφ. σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ παρακαλώ. Ζαν εντάξει. Στη σελίδα 4 είμαστε. Πρώτο τμήμα. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Μετά G. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική H υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε τώρα στην τροπολογία... Α, όχι, δεν θα ψηφίσουμε. Κατά πίπτη αυτή. 258. 260. Υπέρ παρακαλώ. 260 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική I υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική J υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική K, κάπα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική L, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική M, μη υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική N, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική όμικρον, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 33 με προφορική τροποποίηση. Προφορική τροποποίηση πρώτα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα την τροποποιημένη τροπολογία υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική π υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική Q υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική, ο, συγγνώμη, 38, τροπολή 38 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική R υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική S υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 360 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 361 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 362 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική T, τάφ υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική U υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική V υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. της Τζούρι 28 τώρα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική W υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 45 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική X ε, δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ παρακαλώ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική Y τώρα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 50 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική Z υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Η 54 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 36 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική ΑΑ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική ΑΒ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 399 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 58 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική AC υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 60 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 61. Προφορική τροποποίηση. Πρώτα αυτή υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Και τώρα η τροπομένη τροπολογία υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 62 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 1. Υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 63 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 64 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 65 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 66 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 67 έχει αποσυρθεί. 68 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική AD υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 89 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 1 της ΕΝΒΗ με προφορική τροποποίηση. Πρώτα αυτή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροποποιημένη τροπολογία τώρα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. NV2 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 90 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 91 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 92 έχει καλυφθεί. Η 93 έχει καλυφθεί. 94 επίσης από τη συμβαστική R. Συμβαστική τώρα αε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 100 έχει καλυφθεί. 101 με προφορική τροποποίηση. Πρώτα αυτή υπέρ παρακαλώ κατά αποχές εγκρίνεται. Και τώρα ψηφίζουμε την τροποποιημένη τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 102 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 103 υπέρ κατά για να το ελέγξουμε αυτό παρακαλώ. 103 λέει η πρόεδρος. Ελέγχουμε. Ψηφίσατε όλοι. 22 υπέρ, 19 κατά. Εγκρίνεται. Συμβαστική ΑΕΦ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. AG υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. AH υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. AI υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική AJ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 123 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τζούρι 3 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 124 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. MV3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τζούρι 4 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τζούρι 5 υπέρ. Α, όχι, καταπίπτει αυτή. 125 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τζούρι 6 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά τώρα για το τροποποιημένο κείμενο. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι πέρα τη υποφορίας. 39 υπέρ και καμία ψήφος κατά, μία αποχή. Συγχαρητήρια. Τώρα για το ψήφισμα νομοθετικού περιεχομένου, παρακαλώ, το ίδιο. Ψηφίστε, ψηφίστε. Ψηφίστε. Κάποιος δεν έχει ψηφίσει. 39 υπέρ. Κανείς κατά και μία αποχή πάλι. Σας ευχαριστώ. Μπράβο Αλήν. Καλώς. Και τώρα προχωρούμε. Πρέπει να αλλάξουμε λιγάκι στη γραμματεία. Όλοι έτοιμοι. Ωραία, πάμε. Συμβαστική τροπολογία Α. Ψήφι υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική Β. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική C υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. συμβασκή D υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 13 λίμπε υπέρ κατά άποχες ας την ελέγξουμε γιατί εδώ μπορεί να, υπάρχει αποκλει... να υπάρχουν αποκλίνουσες απόψεις πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται με μία αποχή. Πάμε στην ε, συμβιβαστική ε. Η ψηφιπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, όχι, όχι, όχι. 11 της νομικής όχι, εκπίπτει 16 της λίμπε υπέρ, κατά αποχές δεκτή, 17 λίμπε υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, 12 νομικής υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική F υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική G υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική H υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική I υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τζούρι 1 Μπορούμε να τι πάρουμε όλε μαζί. Όχι, όχι. Καλά, δεν πειράζει. Τι να κάνουμε. Τζούρι 1. Υπέρ κατά αποχές δεκτή. 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 7 υπέρ κατά α, α, αποχές. Να ελέγξουμε την 7. Κάποιος δεν ψηφίζει, κλείνω την ψηφοφορία. 23 υπέρ και 15 κατά είναι σαφέ το αποτέλεσμα. Συμβαστική J υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. K υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική L υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Όχι, έχει εκπέσει. Λίμπε 2, υπέρ. Υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 17, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική M, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. ΛΥΜΠΕ 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Λίμπε 9 υπέρ κατά αποχές. Ας ελέγξουμε τη Λίμπε 9 παρακαλώ. Άλλος ένας να ψηφίσει, κλείνει η ψηφοφορία. 21 υπέρ 19 κατά γίνεται δεκτή. Το κείμενο πως έχει τροποποιηθεί έχει η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Άλλη μία ψήφος. Κάποιος δεν έχει ψηφίσει. Ναι. Εντάξει. 39 καμία ψήφος κατά και μία αποχή. Όπως και πριν και ψηφίζουμε το νομοθετικό κείμενο, νομοθετικό ψήφισμα. Μη φύγετε, μη φύγετε. Έχουμε άλλες δύο ψηφοφορίες. Πατήστε τα κουμπιά σας, άλλες δύο έχουμε. Άλλη μία, εντάξει. 39 υπέρ, κάνεις κατά μία αποχή, πολύ ωραία. Μπράβο Αρλίν, μπράβο Αρλίν. επειδή με συγχαίρουν δεν θέλω να πάρω τους επένους. Οφείλονται οι έπαινοι στους σκιώδεις εισηγητές οι οποίοι έχουν κάνει το μεγαλύτερο μέρος της δουλειάς. Και ευχαριστώ και τα μέλη της γραμματείας που έχουν παίξει ένα σημαντικό ρόλο. Ευχαριστώ πολύ. Η εισηγήτρια είναι έτοιμη να μπει σε διαπραγματεύσεις για να διερευνήσει τη δυνατότητα μιας συμφωνίας πρώτης ανάγνωσης για το θέμα αυτό βάσει τη κειμένη διαδικασία η ομάδα διαπραγματεύσεων θα συμπεριλαμβάνει την πρόεδρο, την εισηγήτρια και του σκιώδει. Και η εντολή θα είναι αυτό το οποίο ψηφίσαμε μόλι τώρα, πριν λίγο. Θα επανέλθουμε λοιπόν για την πρόεδρο, για την πρόεδρο των διαπραγματεύσεων. Θα χρειαστεί όμως ένας μήνας περίπου μέχρι να φτάσουμε στους τριγωνικούς διαλόγου. το λόγο. Θεωρώ προσωπικά, λέει ο κ. Γκέμπελς, ότι είναι ένα λάθος. Θα πρέπει πρώτα να πάμε στην Ολομέλεια και να ψηφίσουμε το κείμενο και να μην ψηφίσουμε το νομοθετικό κείμενο και μετά να συζητήσουμε με το Συμβούλιο. Δεν είναι δημοκρατικός ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα αυτά θα πρέπει να σεβαστούμε το δικαίωμα κάθε βουλευτή να καταθέσει τροπολογίες εφόσον το επιθυμούν. Αν πάμε κατευθείαν στις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο, θα καταλήξουμε σε μία συμβαστική λύση που δεν έχουν οι συνάδελφοι τη δυνατότητα να επηρεάσουν. Για λόγους αρχής εγώ είμαι εναντίον της ε, αντιμετώπισης που είχαμε εδώ. Ευχαριστώ, Ρομπέρ. Στην Επιτροπή μας χρησιμοποίησαμε πολλές φορές αυτήν την διαδικασία την, ε, ε, του ελιγμού αυτού να ασκήσουμε πίεση με το να πάμε στην Ολομέλεια πρωτού περάσουμε στον τριμερή διάλογο. Κατανοώ αυτά τα οποία λες, αλλά πιστεύω και η άλλη τεχνική είναι πάρα πολύ χρήσιμη να την έχουμε στο μυαλό μας. Αν, αν δεν υπάρχει κάποια ε, εξέγερση κατά της διαδικασίας που πρότεινα για τις διαπραγματεύσεις, νομίζω ότι γίνεται δεκτή. Κόριν, θες να πεις κάτι εσύ? Νομίζω το επιχείρημα δεν είναι μονάχα το πώς θα ασκήσουμε πίεση, αλλά και το πώς θα μπορούμε να έχουμε μια πιο ισχυρή εντολή από την Ολομέλεια. Νομίζω θα ήταν θετικό να πάμε στην Ολομέλεια, εκτός αν χωρούν αντικειμενικοί λόγοι, να μην πάμε στην Ολομέλεια. Δεν μπορώ να φανταστώ όμως να συμβαίνει κάτι τέτοιο. «39-0» νομίζω ότι είναι μια μεγάλη πλειοψηφία. Είναι μια στεναρή εντολή. Η εισηγήτρια είπε ότι προτιμάει να διαπραγματευτεί. Ναι, θέλετε να πείτε κάτι. Ναι, ναι, θέλω να πω κάτι. Καταλαβαίνω αυτό που λέει ο Ρομπέρ. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου είμαστε σε σύγκρουση, αλλά για το συγκεκριμένο αυτό θέμα είχαμε πολλές συζητήσεις και με τον Επίτροπο Μπαρνιέ. Είχαμε μια μεγάλη ακρόαση, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο έχει κάποια σημασία, διότι προσπαθούμε να κλείσουμε κάποια παραθυράκια τα οποία μας ζήτησε η Κομισιόν να επιταχύνουμε το έργο μας για τα θέματα αυτά. Δεν παραχωρούμε τίποτα. Η δυσκολία, όπως ξέρετε, είναι ότι πρέπει να βρούμε χρόνο στην μέση διάταξη τη Ολομέλεια. Αν θεωρούσα ότι το θέμα αυτό είναι αμφιλεγόμενο, θα έλεγα να πάμε στην Ολομέλεια. Δεν είναι αμφιλεγόμενο και πιστεύω ότι έχουμε καταφέρει να επιταχύνουμε τη διαδικασία για τι διαπραγματεύσει και είναι το πλεονέκτημα δικό μα γιατί το Συμβούλιο έχει καθυστερήσει. Οπότε το Κοινοβούλιο έχει τη δυνατότητα να καθορίσει την μέση διάταξη. Αν περιμένουμε την Ολομέλεια θα καθυστερήσουμε και θα είναι πολύ αργά. Συμφωνώ καταρχήν με τον Ροβέρτο αλλά πρέπει να εφαρμόσουμε αυτό το κανόνα με ευελιξία, ώστε να βγαίνει κάποιο πλεονέκτημα για το Κοινοβούλιο. Ωραία. Εντάξει. Ναι. Δύο διαφορετικά θέματα, λέει ο Ένα θεωρά την τρέχουσα έκθεση και υπάρχει το γενικότερο θέμα που έθεσε ο Ρόμπερτ. Εγώ νομίζω ότι το γενικό θέμα πρέπει να το συζητήσουμε πιο ενδελεχώς. Αλλά εγώ δεν είδα να υπάρχει κάποια αντίρρηση για την τρέχουσα συγκεκριμένη έκθεση, γιατί πρέπει να πάει προηγουμένως στην Ολομέλεια. Ξέρω ότι υπήρξε σε πολλέ επιτροπέ μια συζήτηση για τα θέματα αυτά. Πιστεύω όμως προσωπικά ότι όταν έχουμε πάει με τεχνικές εκθέσεις είχαμε πολύ λίγες τροπολογίες. Συνήθως η πρόταση της Επιτροπής ΕΚΟΝ πηγαίνει στην Ολομέλεια χωρίς αλλαγές. Γιατί αν συμφωνήσουμε εμείς θεωρεί ο κόσμος ότι έχουμε κάποιο κύρος για τα θέματα αυτά και χάρη στο έργο της εισηγήτριας ισχύει και για την τρέχουσα έκθεση. Δεν βλέπω κανένα λόγο σχετικά να δώσουμε καν το μήνυμα ότι κάτι δεν πάει καλά με την έκθεση. Δεν βλέπω λοιπόν ότι ενισχύει την έκθεση το να πάμε στην Ολομέλεια. Είναι περισσότερο μια καθυστέρηση και προτείνω να υπάρξει μια συζήτηση γενικά για τα θέματα αυτά καταρχήν μεταξύ των συντονιστών και μετά στην Επιτροπή μας γιατί το επιχείρημα του Ρόμπετ είναι ένα επιχείρημα γενικής ισχύω γιατί την τρέχουσα όμως έκθεση δεν βλέπω κανένα λόγο να αλλάξουμε τη διαδικασία. Αυτά. Ευχαριστώ. Θα συμφωνώ με τον Ρομπέρτ για αυτά τα οποία είπατε. θα πρέπει να το συζητήσουμε στην Ολομέλεια, στην πρώτη Ολομέλεια. Και αυτό θα πρέπει να ισχύει για τις περισσότερες από τις περιπτώσεις. Στα πλαίσια των επαφών που είχαμε με τις πολιτικές ομάδες και την Επιτροπή, θεωρήσαμε ότι η περίπτωση αυτή δεν είναι ιδιαίτερα προβληματική και υπάρχει μεγάλη συνένεση γύρω από τις προτινόμενες αλλαγές δεν υπάρχουν μεγάλες εκκρεμότητες οι οποίες να τύχουν διαπραγματευτικών προσπάθειών, αλλαγών στην Ολομέλεια. Ακόμα και με το Συμβούλιο τα προβλήματα δεν είναι πάρα πολύ μεγάλα. Για τεχνικούς λόγους λοιπόν μπορούμε να επιταχύνουμε τη διαδικασία. Αλλά βέβαια θα παρακολουθήσω τις απόψεις, τις συζητήσεις. Ίσως θα πρέπει να κάνουμε μια συζήτηση με τους συντονιστές και να προσπαθήσουμε να δούμε ποια θα είναι τελικά η άποψη. Δεν νομίζω ότι το κάθε μέλος πρέπει να πάρει το λόγο πάνω για το συγκεκριμένο. Εγώ λέει Σοφή, συμφωνώ με την πρόταση της Αλήν. Καλώς. Κατανοώ το ότι μπορεί να υπάρχουν διαφορές μεταξύ μας. Κατανοώ και αυτό το οποίο είπε ο Ρομπέρ αλλά αυτό που πετύχαμε στο πακέτο για την εποπτεία, αν δεν ψηφίσουμε και το θέμα της επιβολής, τότε θα υπάρξουν πολλές καθυστερήσεις. Καταλαβαίνετε ότι δεν έχουμε πάρα πολλά μέσα στη διάθεσή μας για να ασκήσουμε πιέσεις. Έχουμε στη συγκεκριμένη περίπτωση ένα θα έλεγα αξιόλογο μέσο, και θα πρέπει να προχωρήσουμε. Τώρα, αν μπορούμε δις να το συζητήσουμε στην Ολομέλεια, δηλαδή ε, στην επομένη αλλά και αργότερα αν χρειαστεί, αυτό θα μας ικανοποιήσει και εμένα και τον κύριο Ρόμπερτ και ο κύριος Ρόμπερτ θα είναι ε, ικανοποιημένος για τον δημοκρατικό τρόπο με τον οποίο θα συζητήσουμε και εγώ θα είμαι ικανοποιημένη λόγω των αποτελεσμάτων που θα έχουμε πετύχει. Μάρκος. Δεν θέλω και εγώ να επιμικίνω τη διαδικασία, αλλά νομίζω ότι όταν έχουμε κάποιες δομές τις ακολουθούμε. Πρέπει να ακολουθήσουμε αυτό το οποίο ψηφίσαμε. Γιατί να μην πάμε. Πιστεύω <clears throat> εγώ ότι είναι καλύτερα να πάμε στην Ολομέλεια γιατί αυτό θα δώσει στους, στους συναδέλφους τα, την, θα τους δώσει τη δυνατότητα να συμβάλλουν στο θέμα αυτό. Είναι ένα θέμα σημαντικό, όπως ήταν το θέμα της Μύφη με την οποία πήγαμε στην Ολομέλεια και δεν υπήρξε κανείς ο οποίος να έχει αντίρρηση τότε όταν πήγαμε στην Ολομέλεια. Συνεχίζουμε τη συζήτηση. Η Ελίζα. Ναι, γιατί σηκώνουν τα χέρια τους όλοι. Υποστηρίζω τη θέση της Αλήν και δεν νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε μια έξι εξαίρεση για το θέμα αυτό. Αλλά σύμφωνα και με τον Ρόμπερτ καταρχήν, δηλαδή νομίζω ότι θα πρέπει να συζητήσουμε και γενικά τι θα κάνουμε. Εγώ συμφωνώ καταρχήν με τον Ρόμπερτ, στη συγκεκριμένη περίπτωση όμως δεν υπάρχει κάποιος λόγος για τον οποίο πρέπει να ακολουθήσουμε την πρακτική που έχουμε ακολουθήσει μέχρι τώρα γιατί υπάρχει και το στοιχείο του κατεπήγοντος. Ο Ούντο, προτού έχουμε μια γενική ρύθμιση, εγώ θα πρότεινα, επειδή καταλαβαίνω και τις δύο πλευρές, θα ήθελα να προτείνω να ακολουθήσουμε το χαμηλότερο κοινό παρονομαστή. Τι θα σήμαινε αυτό. Όσο εσείς ως πρόεδρος μπορείτε να δείτε ότι υπάρχει ένας βαθμός Διαφωνία μεταξύ μα, τότε να πηγαίνουμε στην Ολομέλεια. Αν και η κόρη δεχτεί αυτή την ιδέα, γιατί ζήτησε την ενίσχυση τη θέση που θα έχουμε ως Επιτροπή όπως είναι και στη συζήτηση για το εξάπτυχο. Εγώ θα δεχόμουν λοιπόν αυτό τον κοινό παρονομαστή, εφόσον η πρόεδρο θεωρεί ότι υπάρχει λόγος να πάμε στην Ολομέλεια, τότε να το κάνουμε. Γιατί ο Ρόμπερτ έχει δίκιο. Μερικέ φορές είναι καλύτερο να πηγαίνουμε πράγματι στην Ολομέλεια. Θα κάνουμε λοιπόν ό,τι θέλει ο εισηγητής. Έχουμε ήδη κάνουμε τις ε, απαραίτητες προσαρμογές μεταξύ της έκθεσης της Αρλίν και του Μάρκους. Και έχουμε τώρα διαπραγμάτευση σε δύο διαφορετικούς τριμερείς διαλόγους. Η επόμενη ψηφοφορία τώρα έχει να κάνει με το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο για τον Συντονισμό των Οικονομικών Πολιτικών. Um, Πρώτα απ' όλα, έχουμε μια προφορική τροπολογία, προφορική τροπολογία για τη συμβιβαστική α, ψήφι πέρ. κατά. Αποχές. Γίνεται, απορρίπτεται προφορική τροπολογία, συμβαστική α, υπέρ, κατά. Αποχές Δεκτή. Τροπολογία 15. Υπέρ. Κατά αποχές. Δεκτή. Εκπίπτει τη ΑΦΚΟ 16 ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική Β υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία στη συμβαστική Σ υπέρ κατά απόχες απορρίπτεται. Συμβαστική C. Έλεγχος για την προφορική τροποποίηση στη συμβαστική C. Ηλεκτρονικά. Μόνο η προφορική τροπολογία είναι αυτό που ψηφίζουμε. Ψηφίσατε όλοι. Κλείνω. Απέριπτε. 17 υπέρ 24 κατά. Εντάξει. Πρέπει να ξέρετε τώρα ότι συνήθως βλέπω καλά. Συμβαστική C, υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 28, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 29, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική D, υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 36, υπέρ, κατά, μια στιγμή. 36 και πάλι. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 37. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 38. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική ε. Ε. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Απασχόληση κάτι λέει. Στην παράφορα 24 λέει πρόεδρος στην παράγραφο 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Κάθε μέρος της γραμματείας έχει τη δική του αριθμή. Συμβαστική G υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική H υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τροπορι... Προφορική τροποποίηση στην τροπολογία 51 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 51 ως τροποποιήθηκε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 51, την είπαμε, ναι. Πάμε στη συμβαστική I. Συμβαστική I υπέρ κατά. Πέσαν αυτές οι τροπολογίες, εξέπεσαν, κατέπεσαν, έπεσαν. Συμβιβαστική I λέει το κείμενο. Εντάξει. Έτσι λέει. Συμβιβαστική ΆΗ. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. Γιατί λέει η τροπολογία 54 εδώ, αναρωτιέται η πρόεδρος. Υπάρχει λάθος εδώ. Λοιπόν, απασχόληση παράγραφος 22. Ποιοι είναι υπέρ, κατά. Αποχές, απορρίπτεται. 54 υπέρ. Κατά αποχές, απορρίπτεται. 55 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτό. 56 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Α, έχουμε μία προφορική τροπολογία στην 57. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Θέλετε να υπάρξει ηλεκτρονικός έλεγχος για την προφορική τροπολογία στην 57 παρακαλώ. Ψηφίζετε. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα στις ψηφοφορίες. Δεκτή 22 υπέρ 17 κατά. Περνάμε τώρα στην τροπολογημένη 57. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 57. Ψηφίζεται. Ψηφίζουμε την 57 παρακαλώ. Λοιπόν, δεν έχει γίνει δεκτή η τροπολογημένη τροπολογία. Περνάμε τώρα στην 59. Πρώτο τμήμα ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Υπάρχει μια σύγχυση. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά το πρώτο τμήμα της 59. Εδώ κάποιοι στη μέση δεν ψηφίζουν. Λοιπόν, πείτε μου πώς θα πρέπει να ψηφίσω και εγώ, μη με ξεχνάτε, λέει η Πρόεδρος. Λοιπόν, δεν γίνεται δεκτή. 20 υπέρ και 20 κατά. Το δεύτερο τμήμα λοιπόν, ως έχει τις 59. Ψηφίζουμε το δεύτερο τμήμα τις 59, ηλεκτρονικά. Α, δεν έχει βέβαια νόημα να ψηφίσουμε το δεύτερο τμήμα, λέει τώρα η Πρόεδρος. Ε, θα πρέπει να βγάλουμε τις τρεις πρώτες λέξεις στα αγγλικά. Να ξεκινάει με τη λέξη recommendations, συστάσεις. Ψηφίζουμε το δεύτερο τμήμα λοιπόν. Αν δεν σας αρέσει καταψηφίστε το. Λοιπόν, άλλοι τρεις πρέπει να ψηφίσουν. Ένας από αυτούς είμαι εγώ. Λοιπόν, 25 κατά, 15 υπέρ. Τροπολογία 60. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 61 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική J υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Περνάμε τώρα στην προϋπολογισμός 3. Παράγραφος 3 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 63 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική και η αγγλικό. Ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές δεκτή. Περνάμε τώρα στην 71. Ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 72 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 73 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 74 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 75 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 76 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστική L αγγλικό υπέρ κατά αποχές δεκτό 81 υπέρ κατά αποχές δεκτή προφορική τροπολογία στην συμβιβαστική M από τους φιλελευθέρους υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος παρακαλώ στην προφορική τροπολογία της ALDE για το συμβιβαστικό M αγγλικό 19 υπέρ 21 κατά τώρα έχουμε την προφορική τροπολογία των πρασίνων ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 1 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα, ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, σε δεκτό. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές. Δεν ξέρω αν απερίφθη, αλλά θα πρέπει να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Λοιπόν, ψηφίζουμε τώρα το δεύτερο τμήμα της συμβιβαστικής μη Πέρα της ψηφοφορίας γίνεται δεκτό το δεύτερο τμήμα, 20 υπέρ 19 κατά. Συμβιβαστική λοιπόν εν υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική O υπέρ κατά αποχές δεκτή. 93 υπέρ. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβιβαστική πι αγγλικό υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Πηγαίνουμε τώρα στην 32 της απασχόλησης υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Αύκο 6 υπέρ, κατά, αποχές, Αποχές. Δεν καταλαβαίνω τι γίνεται στο κέντρο της Είναι συνεπώς ελέγχουμε ηλεκτρονικά την 6 της ΑΦΚΟ. Αν δεν ψηφίζετε δεν μπορώ να καταλάβω, λέει η πρόεδρος. Πέρα στις 20 υπέρ, 19 κατά. Καλό ήταν που ελέγξαμε. Λοιπόν, ΑΦΚΟ 4 υπέρ, κατά. Πάλι ηλεκτρονικός έλεγχος για την ΑΦΚΟ 4. Οι φιλελεύθεροι θα πρέπει εν πάση περιπτώσει να σηκώνετε λίγο τα χέρια σας για να καταλαβαίνω τι λέτε. Λοιπόν, ΑΦΚΟ 4 ψηφίζουμε, λέει η Πρόεδρος, ηλεκτρονικά. Πέρα της ψηφοφορίας. Ένας δεν ψηφίζει. 23 υπέρ 16 κατά. Αυκό 5 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 101 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 103 υπέρ. Κατά. Εδώ υπάρχει μια σύγχυση. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για την 103. Υπάρχουν διαιρέσεις στις ομάδες. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική Q υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Αύκο 9 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 107 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Αύκο 19 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Συμβιβαστική R αγγλικά υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Συμβιβαστική S υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 114 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. wasn't adopted. So employment 34 we vote. Employment 34. Λοιπόν, απασχόληση 34 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβιβαστική τι αγγλικό. Τι έγινε με την 114. Υπήρξε ηλεκτρονικός έλεγχος και απερίφθη. Ψηφίζουμε τώρα λοιπόν την 34, απερίφθηκε αυτή με τις ίδιες πλειοψηφίες. Συμβιβαστική τι αγγλικό υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 116 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 117 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Απασχόληση 30 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική U υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική V υπέρ κατά αποχές δεκτή. Απασχόληση 6 είναι υπέρ κατά Αποχές. Απορρίπτεται. Απασχόληση 10 υπέρ κατά. Αποχές. Δεκτή. Απασχόληση 16 υπέρ κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Απασχόληση 23 υπέρ κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Απασχόληση 27 υπέρ κατά Αποχές. Απορρίπτεται. Απασχόληση 33 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Απασχόληση 36 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ινκο 3 λοιπόν υπέρ κατά αποχές δεκτή, Ινκο 4 υπέρ κατά αποχές δεκτή, Ινκο 5 υπέρ κατά αποχές. Νομίζω ότι απορρίπτεται. Ινκο 5 ήταν αυτή. Ψηφίσατε πέρα στις ψηφοφορίες εγκρίνεται. 19-18 το αποτέλεσμα. Ήμκο 6 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Ήμκο 7 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Ήμκο 8 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Ήμκο 9 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Ήμκο 10 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Ήμκο 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. άφκο 2 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. άφκο 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. άφκο 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Θέλετε να το ελέγξω, γιατί ήταν οριακό. Αύκο 13. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα της ψηφοφορίας. 23 υπέρ, 14 κατά είναι σαφές τελικά. 14 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Αύκο 15 υπέρ, κατά, αποχές θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά και την 15, γιατί και αυτό είναι οριακό το αποτέλεσμα. Ψηφίσατε όλοι. Τώρα ακόμα. Δεν ψηφίζετε, ωραία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 18 υπέρ, 19 κατά. Απορρίπτεται. Αύκο 18 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται, αλλά θέλω να το ελέγξουμε και αυτό. Ψηφίσατε όλοι, πέρας της φοφορίας. Απορρίπτεται. 16 υπέρ, 22 κατά. Αύκο 20 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Γυναίκες, πρώτη υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Φεμ 2 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Φεμ 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Φεμ 4 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Φεμ 5 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Φεμ 6 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Φεμ 7 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Φεμ 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Φεμ 9 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Φεμ 10 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Φεμ 11 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Φεμ 12 υπέρ κατά αποχές σύγχυση. Θα ελέγξουμε για την ΦΕΜ 12. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας τις φοφορίες. Πέρας. 18 υπέρ, 20 κατά. Απορρίπτεται. Αιτιολογικές σκέψεις τώρα. Τροπολογία 4 υπέρ. Κατά. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας της ψηφοφορίας. 19-19 απορρίπτεται. Οπότε αρχικό κείμενο στην ατολική σκέψη α υπέρ παρακαλώ, κατά αποχές εγκρίνεται. 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Αρχικό κείμενο όχι. 7. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 8. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 9. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Απασχόλησης α υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Απασχόληση β υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Σ δεν ψηφίζουμε. Δέλτα, δι υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Έψιλον ε απασχόλησης υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τα επόμενα όχι. Πάμε στην ΙΜΚΟ ΑΕ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Γυναικών Ε υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Β γυναικών υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Γυναικών Σ υπέρ κατά αποχές Απορρίπτεται. Ετιολογικέ αναφορέ τώρα. 1. Υπέρ. Κατά. αποχέ, Εγκρίνεται. 2. Υπέρ. Κατά. αποχέ, Εγκρίνεται. Τι θέλετε. Όλε αυτέ μαζί. πόσε είναι. Ετιολογικέ αναφορές μέχρι και τη 10. Υπέρ, κατά, απόχέ. Ωραία, εγκρίνονται όλες. Τώρα, προφορική τροπολογία του συγγετή υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τώρα, τι κάνουμε. Τις ψηφίσαμε όλες έτσι, σωστά. Αιτιολογική σκέψη, μάλλον αναφορά 39. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Αρχικό κείμενο υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Υμκο... 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ήμκο 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα το τροποποιημένο κείμενο παρακαλώ με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ψηφίστε. Ψηφίσατε όλοι. πέρα τη ψηφοφορίας. 30 υπέρ, 8 κατά και καμία αποχή. Σας ευχαριστώ πολύ. Πέρας τη ψηφοφορίας. Τώρα, σας ευχαριστώ πολύ όλους. Ο Πάντλο θα αναλάβει την Προεδρία τώρα για το τελευταίο σημείο που έχουμε στην ημερήσια διάταξη. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα περάσουμε τώρα στο επόμενο θέμα. Με εισηγητή τον Αφρέντο Παλώνε για τα δημόσια οικονομικά στην ΟΝΑ. για το 2011 και για το 2012. Θα δώσω το λόγο λοιπόν στον κύριο Παλώνε. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα είμαι σύντομος γιατί πολλοί από τους συναδέλφους έχουν κουραστεί και μπορούν έτσι και αλλιώς να διαβάσουν αυτό το σχέδιο έκθεσης. Εγώ έχω διαιρέσει το πρόγραμμα αυτό για, την, το δημοσιονομικό κομμάτι της ΟΝΕ σε τέσσερα αν θέλετε σημαντικά τμήματα. Τέσσερα τμήματα που αφορούν τη σημερινή κατάσταση, τις διαφορές ανάμεσα στις χώρες, στην ενίσχυση των προϋπολογισμών και τέλος στην σημασία που έχει η ανάπτυξη που είναι θα έλεγα το βασικό θέμα έτσι όπως παρουσιάζονται τα πράγματα σήμερα. Είδα ότι υπάρχουν διαφορές ανταγωνιστικότητας και προβλήματα στα δημοσιονομικά ανάμεσα στις χώρες και αυτά δημιουργούν προβλήματα στην οικονομική ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο σύνολό της. Η οικονομική διακυβέρνηση μέσω του εξαπλού πακέτου και του τετραπλού πακέτου και με το δημοσιονομικό σύμφωνο βλέπουμε ότι υπάρχει η δυνατότητα να γίνουν σημαντικά βήματα προς τα εμπρός στον οικονομικό τομέα, αλλά αυτό δεν αρκεί. Έχουμε βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και νομίζω έχουμε θέσει και στόχους δημοσιονομικούς οι οποίοι ναι μεν είναι πολύ ενδιαφέροντες αλλά από μόνοι τους δεν είναι κάτι το οποίο αρκεί. βλέπουμε ότι υπάρχουν πολύ σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις χώρες και σε επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης και σε επίπεδο σταθεροποίησης των δημοσιονομικών. Υπάρχει μια σαφής διαφοροποίηση ανάμεσα στους πιλότους του Βορρά, στους ε, ε, θα έλεγα χώρες που πρωτοπορούν στον Βορρά και στις χώρες του Νότου. Υπάρχουν προβλήματα λόγω της γραφειοκρατίας τα οποία ισχύει σε ορισμένες χώρες, λόγω του κλίματος του ευνοϊκού για τις επιχειρήσεις σε ορισμένες χώρες και του μη ευνοϊκού σε κάποιες άλλες. Νομίζω ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές και για πάρα πολλούς λόγους τελικά υπάρχουν οι διαφορές αυτές και γι' αυτό απαιτούνται διαφοροποιήσιμες στρατηγικές από τη μία χώρα στην άλλη. Να εξηγηθώ. Οι συστάσεις ε, τις οποίες έχει εκδώσει το Συμβούλιο στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου δεν μπορεί να είναι ταυτόσιμες για όλες τις χώρες, γιατί αντικειμενικά οι συνθήκες που σοφούν σε κάθε χώρα είναι διαφορετικές. Υπάρχουν ε, χώρες οι οποίες ε, απαιτούν ιδιαίτερες προσπάθειες, εντατικές προσπάθειες και άλλες λιγότερο. Σε κάποιες χώρες απαιτούνται διαφορετικές ε, θα έλεγα παρεμβάσεις, ε, ιδιαίτερα στις χώρες με υψηλότατο δημόσιο χρέος. Και όταν ε, αναφερόμαστε στην σταθεροποίηση των δημοσιονομικών και την εξυγίανση των δημοσιονομικών, πρέπει να υπάρξει μια ισορροπία στα δημόσια οικονομικά της χώρας, η οποία θα βοηθήσει την ανάπτυξη της απασχόλησης. Γίνεται μια συζήτηση γύρω από το θέμα αυτό, και δεν κρύβω ότι και η δική μου χώρα είναι κάτι το οποίο φυσικά με απασχολεί. Είναι μια χώρα η οποία ίσως έζησε άνω των δυνατοτήτων της, επιβαρύνοντας και μεταφέροντας τις μελλοντικέ σε το θέμα του δημόσιου χρέους, το οποίο θα ονόμαζα, θα έλεγα, χρέος γενεάς ουσιαστικά. Θα πρέπει λοιπόν να γίνουν περισσότερες προσπάθειες για την εξυγίαση των δημοσιονομικών και θα πρέπει να γίνουν ακόμα και περισσότερες. Οι προσπάθειες έχουν ξεκινήσει βέβαια, επαναλαμβάνω ότι πολλές είναι οι χώρες στην ε, περιφέρεια της Ευρώπης που κάνουν τεράστιες προσπάθειες. Θα πρέπει όμως να διευκρινίσουμε ακόμα καλύτερα το εξής. Η εξυγίανση των οικονομικών θα πρέπει να βασιστεί κυρίως και στην δημόσια δαπάνη, στις δημόσιες επενδύσεις. Είμαι πεπισμένος γι' αυτό και όχι μόνο σε σχέση με την αύξηση των εσόδων. Αν μείνουμε σε αυτό το οποίο προτείνω, αποφεύγουμε εν πολύ στον κίνδυνο της ύφεση και θα μπορέσουμε να ενεργοποιήσουμε την ανάπτυξη μεσοπρόθεσμα. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να αποφύγουμε λοιπόν να πιέσουμε μονομερός φορολογικά. Γιατί αυτό θα αυξήσει το κόστος της εργασίας, θα αυξήσει το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων και θα οδηγήσει σε μειώσεις, αν θέλετε, του κόστους λειτουργίας συνολικά των επιχειρήσεων εις βάρος των δραστηριοτήτων τους. Λοιπόν, Σχετικά με το δημόσιο χρέος, θα ήθελα να διευκρινίσω την εξής άποψη. Τα μέτρα λιτότητας από μόνα τους δεν κάνουν τίποτα. Θα πρέπει να συνοδεύονται από μέτρα δικαιοσύνης στον τομέα των φορολογικό και θα πρέπει αυτά τα μέτρα να μην οδηγήσουν στην μεγαλύτερη ύφεση, να μην οδηγήσουν σε ένα φαύλο κύκλο στον οποίο αν ξεκινήσουμε και μπούμε οι μειώσεις και οι περικοπές δεν θα είναι ποτέ αρκετές χωρίς δογματισμούς αλλά με απαρκή ρεαλισμό εάν δεν υπάρξει οικονομικός ρεαλισμός δεν θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε μια πραγματική δημοσιονομική εξυγίανση. Το να μειώνουμε τις δημόσιες δαπάνες είναι κάτι το οποίο δεν οδηγεί συνεχώς πουθενά. Ευχαριστώ κύριε Παλώνε. Οι σκιώδεις ε, έχουν το λόγο τώρα για τη σοσιαλιστική ομάδα, ο κύριος Χουαν Κόγκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον εισηγητή για το σχέδιο εκθεσής του. Είναι πάρα πολύ σύντομο, είναι λίγες σελίδες και αντίθετα <clears throat> από ό,τι ανέφερε ο ίδιος έχει μια δογματικότητα στην αναλύση των πολιτικών προϋπολογισμού. Εδώ είναι και ο πυρήνας της πολιτικής και οικονομικής συζήτησης. Δηλαδή, ποια θα πρέπει να είναι η πολιτική, η δημοσιονομική, με την οποία να αντιμετωπίσουμε την ύφεση η οποία έχει εγκατασταθεί στην Ευρώπη. Σχετικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να εκφράσει την άποψή του για δύο εκθέσεις. Έχει εκφράσει ήδη τη θέση του πέρσι και φέτος. Αλλά έκτοτε έχει αλλάξει το πλαίσιο. Αν το Σεπτέμβριο του 2011 θεωρούσαμε ότι τα μέτρα λιτότητος και η εξυγίανση θα οδηγούσαν σε οικονομική ανάκαμψη βάσει των δικτών της, επι... της εποχής εκείνης, σήμερα αυτή είναι μια άποψη που είναι πολύ δύσκολα να, δύσκολα την υποστηρίξει κανείς. Έχουμε ανεργία 11,5 σχεδόν 100 κατά μεσονόρο. Είμαστε το 0,2% κατά μέσον όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση το δεύτερο εξάμεινο του 2012 και παρόλα αυτά οι κυβερνήσεις έχουν κάνει όλα αυτά τα οποία τους ζητήθηκαν τα τελευταία δύο χρόνια. Και δυστυχώς η έκθεση της Κομισιόν περιορίζεται στο να διαπιστώσει, όπως παραθέτω, ότι η ευρωπαϊκή οικονομία δεν εξεπλήρωσε τις ελπίδες που είχαμε θρέψει πέρσι όταν εξεδόθη αυτή η έκθεση η Κομισιόν δεν κατανοεί και δεν μπορεί να αποδεχθεί ότι η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε απέτυχε. Αν ίσχυαν όλα αυτά που λέει η Κομισιόν θα μειωνόταν η ανεργία και η Ελλάδα θα ήταν από τις πιο ανταγωνιστικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει. Μπορούμε να συζητήσουμε για τη διάγνωση που κάνετε και για την οποία επιμείνατε στην παρουσίασή σας. Μήπως επειδή έχουμε δαπανίσει υπερβολικά έχουν αυξηθεί τα ελλείμματα ή γιατί στις περισσότερες χώρες έχουμε μειώσει τους φόρους. Αν δείτε τι έχει γίνει τα τελευταία δέκα χρόνια, οι περισσότερες χώρες έχουν συγκρατήσει τις δαπάνες τους, αλλά έχουν μειωθεί τα φορολογικά έσοδα, όχι μονάχα γιατί έχουν μειωθεί οι φόροι, αλλά γιατί και αυτές οι πολιτικές μείωσης των φόρων δεν είχαν τα προσδοκόμενα αποτελέσματα σε σχέση με την αύξηση της οικονομικής μεγέθυνσης. Εσείς λέτε και ο ίδιος σε μία φράση ότι για τις δαπάνες δεν θα πρέπει να περικόψουμε τις δαπάνες δημοσίων επενδύσεων και εφιστώ την προσοχή σας σε ένα λάθος πολύ ενδιαφέρον στη γαλλική μετάφραση όπου λέγεται ότι στο σημείο 9 νομίζω είναι αυτό, στη σελίδα 5. Υπενθυμίζει ότι η σχέση μεταξύ ανάκαμψης και εξυγίανσης λέει ότι η εξυγίανση είναι η μείωση των δαπανών και, η, και όχι η αύξηση των ε, εσόδων. Αυτά λοιπόν λέτε εκεί πέρα. Υπάρχει ένα σφάλμα λοιπόν στη μετάφραση. Εγώ νόμιζα για μια στιγμή ότι υποστήριζε τον Γκέινς. Όχι όμως δυστυχώς. Δεν είναι αυτή η φιλοσοφία δικιά σα. Αυτό ήταν μια υποσημείωση. Σοβαροτέρος. Τον Ιούνιο υπήρξε ένα ορόσημο στην οικονομική συζήτηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί στις διάσκεψει κορυφή 28 και 29 Ιουνίου αναγνωρίστηκε ότι η στρατηγική αυτή θα έπρεπε το λιγότερο να αναθεωρηθεί. Και το σύμφωνο ανάπτυξης, το οποίο συμφωνήθηκε, έδειχνε ότι πρέπει να κινητοποιήσουμε τους πόρους για να υπάρξουν κάποιες δαπάνες για το μέλλον, αναφέρθηκε το ποσό των 120 δισεκατομμυρίων, για να υποστηριχθεί η ανάκαμψη. Έκτοτε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ανακοίνωσε ότι θα παρενέβαινε για να μειώσει την κερδοσκοπία σε σχέση με το κρατικό χρέος. Η Ισπανία και η Πορτογαλία κατάφεραν να έχουν ένα, μια επαναδιαπραγμάτευση του χρονοδιαγράμματος για τη μείωση του έλλειμματός τους, γιατί ξέρουν ότι με την ύφεση δεν θα μπορέσουν να τηρήσουν τις προσίες τους για το 2013. Ο κύριος Μάριο Μόντι από τη χώρα σας την ίδια τόνισε ότι πρέπει να, να εξαιρεθούν οι δημόσιες επενδύσεις από το έλλειμμα, από τον υπολογισμό του πρωτογενούς ελλείμματος, ο κύριος Μοντή πιστεύει πράγματι ότι θα πρέπει να υπάρξει μια τέτοια κίνηση η οποία θα τονώσει τις δημόσιες επενδύσεις, αντίθετα με αυτά που λέει ο ΣΥΓΙΤΙΣ. Το Σύμφωνο λοιπόν Ανάπτυξης επέτρεψε να επιβεβαιώσουμε την επιθυμητή δημοσιονομική εξυγίανση επιβεβαιώνει την ανάγκη να υπάρξει όμως και μια διαφοροποιημένη αντιμετώπιση η οποία προωθεί την ανάπτυξη, ιδίως με την υποστήριξη των επενδύσεων οι οποίες έχουν χαρακτήρα αναπτυξιακό. Λυπάμαι που δεν βλέπω αυτή τη νέα προσέγγιση η οποία είναι υποσυζήτηση σε, ευρωπαϊκή, ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο στο σχέδιο έκθεσή σας το οποίο απλώς επαναλαμβάνει τις ε, ρετσέτες της Κομισιόν οι οποίες μέχρι στιγμής είναι φανερό ότι έχουν αποτύχει και στο παιχνίδι που παίζουμε σήμερα σε θεσμικό επίπεδο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να είναι πιο μπροστά από το Συμβούλιο και βασιζόμαστε στη δική σας ευφυΐα κύριε ε, εισηγητά για να μην υπολοιπόμεθα του Συμβουλίου αλλά να προηγούμεθα αυτού. Ευχαριστώ. Ο κύριος Τρεμόσα από τους ε, φιλελεύθερους. Θα μιλήσω Ιταλικά προς τιμή του κυρίου Παλώνε που προετοίμασε την έκθεση αυτή. Νομίζω ότι θα είναι εύκολο για τους φιλελευθέρους να υποστηρίξουν την έκθεση αυτή γιατί υπάρχουν πάρα πολλά θέματα στα οποία συμφωνούμε. Σαν παράδειγμα, εγώ συμφωνώ ότι ένα τέτοιο είδους προϋπολογισμός είναι προϋπόθεση για την οικονομική ανάκαμψη. Όταν μιλάμε για την Ισπανία σαν παράδειγμα θα δούμε ότι τα τελευταία τέσσερα χρόνια δεν ξεκίνησαν, δεν είχαν ξεκινήσει μέτρα λιτότητας. Συνεχίζουμε με ένα δημόσιο χρέος το οποίο φτάνει το 8,10% του ΑΕΠ τα τελευταία 4 χρόνια. 12, 11, 10 και 9. Λοιπόν, ας μιλήσουμε για, το φαινόμενο crowding out που χώρες ε, που κάνουν τεράστιες προσπάθειες ε, στον τομέα τον γνωρίζουν καλά. Βλέπουμε ότι δεν υπάρχουν ιδιωτικές επενδύσεις, δεν υπάρχουν δυνατότητες επενδυτικές, υπήρξε θα έλεγα μια μείωση του ΑΕΠ στον τομέα των επενδύσεων κάτω του 50%. Δεν μπορούμε λοιπόν να προσελκύσουμε πλέον χρήματα. Αυτά αγαπητές συνάδελφε της σοσιαλιστικές ομάδες ε, υπάρχουν και στον προϋπολογισμό της Ένωσης. Ο Πάρσον ήταν πρωθυπουργό της Σουηδίας στη δεκαετία του 90 και χάρη στα δικά του μέτρα μπορούμε να μιλήσουμε για την λιτότητα σαν προήμιο της ανάκαμψης. Μου είχε πει γιατί έρχεται κάθε μήνα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γίνεται μια συνάντηση για την δασοκομική πολιτική. Και είχε πει ότι την πρώτη φορά που έγινα εγώ πρωθυπουργό μιας σοσιαλδημοκρατική κυβέρνησης μείωσα τη δημόσια δαπάνη κατά 10% του ΑΕΠ. Έκανε μια οριζόντια περικοπή σε όλα τα κεφάλαια των δαπανών για να ανακτήσει έναν ισορροπημένο προϋπολογισμό και δύο χρόνια μετά η χώρα του βγήκε από την οικονομική κρίση. Και σήμερα ο Πάρσον δίνει, δίνει παρουσιάσει σε όλο τον κόσμο για το πώς μπορεί κανείς να ξεφύγει από μια τόσο σοβαρή και επικίνδυνη κρίση. Πρέπει λοιπόν να συνεχίσουμε με μια συζήτηση χωρίς δογματικές αιμονές και εμείς οι φιλελεύθεροι είμαστε θα έλεγα πιστοί σε αυτά τα οποία πιστεύουμε και λέγουμε εδώ εδώ και τρία χρόνια στην Επιτροπή ότι πρέπει να ισορροπηθεί ο προϋπολογισμός εάν θέλουμε να, ανακτήσουμε την ανάπτυξη και την εμπιστοσύνη στις χώρες μας. Με τον κύριο Παλώνε ε, δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω σε πάρα πολλά από αυτά που λέει. Θα πρέπει για να πετύχουμε αυτήν την ισορροπία θα έλεγα να μειώσουμε τις δαπάνες και όχι τόσο να αυξήσουμε τους φόρους. Θα πρέπει να δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα μέσω της αύξησης των περικοπών αλλά όχι της φορολογίας. Ίσως πολλές χώρες να έχουν την δυνατότητα να μειώσουν τη δημόσια δαπάνη σε διάφορες πολιτικές υποδομών σαν παράδειγμα. Απ' την άλλη υπάρχουν επενδύσεις σε ορισμένες χώρες που δεν έχουν πραγματικό νόημα σε σχέση με το κόστος τους. Υπάρχουν ορισμένες χώρες στο νότο της Ευρώπης όπου ακόμα και σήμερα αναπτύσσεται και αυξάνεται ο αριθμός αυτών που εργάζονται ε, στον δημόσιο τομέα. Γνώμη μας είναι ότι έτσι δεν πάμε πουθενά. Και αυτό το οποίο μου άρεσε ε, ιδιαίτερα στην έκθεση του κυρίου Παλώνε είναι το σημείο 14. Στο σημείο 14 ο κύριος Παλώνε αναφέρεται στα κράτη-μέλη και διευκρινίζει τις ευθύνες των διαφορετικών επιπέδων διακυβέρνησης κεντρικής, περιφερειακής, ευρωπαϊκής αν θέλετε, έτσι ώστε ο καθένας να μπορέσει να κάνει μια προσπάθεια αποκατάστασης της ισορροπίας της δημοσιονομικής. Εγώ σαν καταλανός είμαι ιδιαίτερα ευαίσθητος σε αυτά, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο ε, θα ισχύσει και για τις αποκεντρωμένες σε επίπεδο δημοσίων δαπανών χώρες. Στην ισπανική περίπτωση υπάρχει αυτό που ονομάζουμε ένα blame game, δηλαδή ο καθένας κατηγορεί τον άλλο ε, στα πλαίσια της ε, θα έλεγα προσπάθειας φυγοκεντρικής απαλλαγής από το δημόσιο χρέος, η κυβέρνηση ξαφνικά ανακάλυψε ότι α, δεν φταίμε εμείς, αυτά είναι οι περιφέρειες οι οποίες ε, έχουν λιγότερα έσοδα και περισσότερες δαπάνες. Συμφωνώ λοιπόν με τον εισηγητή για αυτά τα οποία λέγει και νομίζω ότι θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε προς την κατεύθυνση αυτή γρήγορα. Εκ μέρου των Πρασίνων τώρα, ο κύριος Γκυγκόλ έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σύντομα κάποιες παρατηρήσεις. Αντικαθιστώ τον σκιώδη μας, το Σάικαουτ, από τις κάτω χώρες, την κυρία Μποσκάουτ. Αντίστοιχες παρατηρήσεις έχουμε και εμείς να κάνουμε. Πιστεύουμε ότι τα γη δημοσιονομικά είναι το σημαντικό αλλά από την άλλη μεριά έχει μεγάλη σημασία το πώς θα το πετύχουμε, ποια μέθοδο θα ακολουθήσουμε δηλαδή. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα επιτρέψτε μου να σας πω πως πιστεύω ότι η αναφορά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το θέμα αυτό των ε, δημοσιονομικών είναι θετικό, είναι καλό. Εγώ ήμουν εισηγητής για αυτή την υπόθεση στην προηγούμενη έκθεση που κάλυπτε και αυτό το θέμα. Πιστεύουμε λοιπόν ότι ουσιαστικά η έκθεση αυτή πρέπει να είναι πιο λεπτομερής ήδη από το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, γιατί η Επιτροπή έχει επενδύσει μεγάλες προσπάθειες για να αναλύσει σημαντικά θέματα όπως είναι ε, το πολυοπλαστικό φαινόμενο και διάφορες άλλες περιπτώσεις με συγκεκριμένα ποσά. Στην έκθεση ως έχει τώρα δεν είναι ξεκάθαρο το ότι εμείς έχουμε υποχρέωση να αναφέρουμε, να μελετούμε και να σχολιάζουμε την ε, τόσα λέει Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εμείς πρέπει να αναλάβουμε το θεσμικό μας ρόλο και να είμαστε ξεκάθαροι στο σχέδιο κειμένου επ' Δεύτερον, συμφωνώ με τα γενικά που λέει ο εισηγητή, τι βασικές γραμμές για τη σημασία που έχουν τα υγιή δημοσιονομικά, ότι πρέπει να επανέλθει η ισορροπία σε αυτά κλπ. Τα έχουμε δει και ξαναπεί, να μην τα επαναλάβω. Εκεί όμως που διαφωνούμε είναι στο ότι μπορείτε απριόρι να πείτε ότι η εξισορρόπηση πρέπει να γίνεται από πλευρά των δαπανών περισσότερο από ό,τι από πλευρά των εσόδων. Η φορολογική πίεση και οι επιπτώσεις στην αγορά και στην ανάπτυξη ε, είναι κάτι πολύ αμφίβολο γιατί έχετε χώρες που έχουν ψηλή φορολογία, οι βόρειες χώρες για παράδειγμα και είναι οι πιο ευτυχείς χώρες στον κόσμο και έχετε άλλες χώρες οι οποίες έχουν υψηλή φορολόγηση που όμως τίθενται διάφορα ερωτήματα. Για παράδειγμα, στη χώρα που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, αλλά εν πάση περιπτώσει να μην σχολιάσω πάνω σε αυτό. Θέλω να πω ότι δεν αποτελεί βασικό και καθοριστικό στοιχείο το πόσο ψηλή είναι η φορολογία. Το θέμα είναι ποιος την πληρώνει και τι την κάνουμε. Οπότε τα γενικά για το πώς να βγούμε από τα δημοσιονομικά προβλήματα αυτό δεν είναι ένα γενικό σχόλιο που μπορεί να κάνει κανείς. Μερικές φορές είναι προτιμότερο να αυξήσουμε τη φορολογία, άλλες φορές είναι καλύτερο να μειώσουμε τις δαπάνες και άλλες φορές είναι καλύτερο να επενδύσουμε στην ανάπτυξη. Κάθε φορά είναι θέμα πολιτικού μείγματος το τι είναι καλύτερο. Οπότε θα ήμουν πολύ προσεκτικός για τέτοιες δηλώσεις. Επιπλέον εμείς πιστεύουμε ότι εφόσον είναι αναγκαία διαδικασία εξισορρόπησης των δημοσιονομικών των χωρών, και πρέπει να γίνουν προσπάθειες, πρέπει να τηρήσουμε και τους στόχους του 2020. Τα μέτρα δηλαδή δεν θα πρέπει να πλήξουν τους στόχους που έχουμε κρίνει ως αναγκαίους και έχουμε ψηφίσει για το 2020. Γι' αυτό και πιστεύουμε ότι η διατύπωσή μας πρέπει να είναι έντονη. Να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των δημοσιονομικών συγχρόνως να αντιμετωπιστεί η ένδια, να αυξηθεί η απασχόληση, να επενδύσουμε στο μέλλον. Αυτά τα πρέπει να τα λέμε με έντονο ύφος. Θα υποβάλουμε τις τροπολογίες μας και μια που έχουμε συνεργαστεί και κατά το παρελθόν μαζί, σίγουρα θα συνεργαστούμε και πάλι πολύ καλά. Και ας ελπίσουμε ότι θα πετύχουμε να βγάλουμε ένα ισχυρό μήνυμα. Υπάρχει όμως και ένα πρόβλημα μετάφρασης από ότι τα αγγλικά μου δεν είναι μεν πολύ καλά, ίσως, αλλά ελπίζω να με καταλάβατε. Πολύ καλά είναι τα αγγλικά σου, Σβεντάνκεσεν, λέει ο πρόεδρος. Δεν υπάρχει κανείς εδώ ούτε από τη Σιάρου, από την οπότε θα δώσω το λόγο τώρα σε όποιους άλλους ζητάνε το λόγο. Η κυρία Ποδηματά, παρακαλώ κυρία Ποδηματά. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον συγητή για το έργο του και για τα σχόλιά του. Κάποιες παρατηρήσεις για το σημαντικό αυτό θέμα. Από τη δική μου πλευρά, πρώτα απ' όλα να σας υπενθυμίσω ότι επειδή βρισκόμαστε στο μέσο μιας πολύ σοβαρής οικονομικής και κοινωνικής κρίσης πρέπει να διατηρούμε στο πνεύμα μας το γεγονός ότι υπάρχουν κάποια γιατί και κάποια πώς που πρέπει να απαντήσουμε σε σχέση με αυτή την κατάσταση. Τα δημόσια οικονομικά δεν απέτυχαν, δεν αστόχησαν μόνο λόγω εθνικών ευθυνών, Η κρίση η ίδια δεν είναι απόρρια προβλημάτων στα δημόσια των οικονομικά και αστοχιών στα δημόσια οικονομικά. Ναι λοιπόν, πιστεύω τα δημόσια οικονομικά φυσικά παίξανε ρόλο και υπήρξαν σημαντικές εθνικές ευθύνες στον τομέα αυτό που πρέπει να τις αναγνωρίσουμε και να τις πάρουμε στα σοβαρά. και πρέπει να αναλάβουμε και το πολιτικό κόστος αυτής της αναγνώρισης, αλλά συγχρόνως θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι οι αποτυχίες στα δημόσια οικονομικά είναι αποτέλεσμα ενός γενικευμένου συστημικού προβλήματος πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι υπήρξε και υπάρχει σε μεγάλο βαθμό. Μέσα στην Ευρω... Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Το θέμα δεν είναι λοιπόν να βρούμε το γιατί και το πώς. Οδηγηθήκαμε στην τωρινή οικονομική κρίση. Και σίγουρα δεν πρέπει να το κάνουμε αυτό, να κάνουμε μια τέτοια αναζήτηση μόνο σε επίπεδο εθνικό γιατί, και κατακαιρματισμένο, γιατί αυτό μπορεί να μας οδηγήσει σε, λαθασμένες σε συμπεράσματα και λαθασμένες συνταγές για να αντιμετωπίσουμε το θέμα. Αυτό παραμένει η δημοσιονομική εξυγίανση μια αναγκαιότητα και για κοινωνικούς και για οικονομικούς λόγους. Είναι μια προϋπόθεση για την ανάπτυξη, γιατί πάνω απ' όλα είναι απαραίτητη για να επιτευχθεί ένα αποδεκτό επίπεδο βεβαιότητας που θέλει να έχει οποιοδήποτε οικονομικός φορέας για να αγοράζει, να πωλεί, να λειτουργεί σε οποιαδήποτε οικονομία. Συγχρόνως όμως η δημοσιονομική εξυγίανση έχουν δημιουργήσει και ένα φαύλο κύκλο λιτότητος και ύφεσης. Έχουμε χώρες, σαν ο Λίαμ στην Ελλάδα, δεν είναι μονάχα η Ελλάδα, έχουμε την Ιρλανδία, έχουμε την Πορτογαλία, την Ισπανία, έχουμε πολλές χώρες οι οποίες έχουν που έχουν επιμελέστατα εφαρμόσει τα μέτρα τα οποία τους ζητήθηκε να εφαρμοστούν, αλλά παρά τις σοβαρές αυτές περικοπές που επέφεραν τα τελευταία τρία χρόνια, σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό έχουν δει το δυναμικό τους, τη δυνατότητα εξυγένσης να περιορίζεται από την ύφεση για τη χώρα Να σας δώσω ένα μικρό παράδειγμα. Για κάθε 100 ευρώ περικοπών στην Ελλάδα, το φορολογικό χάσμα που καταφέρνει να γεφυρώσει η χώρα μου είναι λιγότερο από 80 ευρώ. Και συγχρόνως πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι μια ανάλυση βιωσιμότητας για οποιοδήποτε οικονομικό εγχείρημα περιλάμβανε τα προγράμματα ιδιωτικοποίησης όπου οι καθυστερήσεις επεκριθήσαν ιδιαίτερα και τα οποία δεν τήρησαν τα κριτήρια για δυνητικούς επενδυτές. Πέραν λοιπόν των οικονομικών προβλημάτων, αντιμετωπίζουμε τώρα κοινωνικά και πολιτικά προβλήματα και αυτό φυσικά ισχύει και για άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα, ανάδυση του ρατσισμού. Έχουμε δείγματα μιας σοβαρής κοινωνικής κρίσης και μαζί πολιτικής και οικονομικής κρίσης και αυτό είναι κάτι που πρέπει να λάβουμε πολύ στα σοβαρά. Εν κατακλείδη λοιπόν, η πρότασή μου θα ήταν, εφόσον πολλές από αυτές τις πτυχές έχουν οδηγήσει σε αναγνώριση της ανάγκης μιας πολιτικής πρωτοβουλίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πιστεύω ότι χρειαζόμαστε να υπογραμμίσουμε πέραν των εθνικών προσεγγίσεων για τα δημόσια οικονομικά, θα πρέπει να υπογραμμίσουμε και μια ευρωπαϊκή προσέγγιση η οποία πέραν των εθνικών υπευθυνοτήτων και απαραίτητων δράσεων που πρέπει να παραμείνουν σε εθνικό επίπεδο βλέπει και τη δυνατότητα να υπάρξει μια ευρωπαϊκή προσέγγιση για να αντιμετωπιστούν και τα δημοσιονομικά προβλήματα και τα προβλήματα οικονομικής ανάπτυξης μέσα σε ένα κοινό πλαίσιο πολιτικών που θα πρέπει να προωθηθούν. Όλα αυτά σημαίνουν μια ολιστική προσέγγιση για την πολιτική του προϋπολογισμού, για την πολιτική πρόθεση της ανάπτυξης και απασχόλησης μέσω κοινών πολιτικών και διαφθορτικών πολιτικών και πρέπει να τις αναδιατυπώσουμε ή να αλλάξουμε τις προτεραιότητές τους. Τι, σημαίνουμε, τι εννοούμε με διαφορετικές αλλαγές και ποιες είναι οι διαφορετικές αλλαγές στις οποίες δίνουμε προτεραιότητα. Αυτό είναι λοιπόν το σημαντικό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κυρία Ποδηματά. Ο εισηγητής τώρα, κύριο Παλών, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Νομίζω ότι η διαλεκτική και η δημοκρατία έχουν μεγάλη σημασία γιατί έτσι μόνο μπορούμε να καταλήξουμε σε ενδιαφέροντες συμβιβασμούς. Υπήρξαν διαφοροποιήσεις, υπήρξαν αντιπαραθέσεις και θα ήθελα να πω στον κύριο Γκίγκολντ. όταν εγώ κάνω μία, θα έλεγα, αναφέρομαι σε μία θέση μου, έστω και προκλητική, αυτό δεν σημαίνει ότι διαφωνούμε σε όλα. Σαν παράδειγμα, στους ε, ε, ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς φυσικά και συμφωνούμε. Όλες οι χώρες θα πρέπει να έχουν προϋπολογισμούς οι οποίοι ε, να είναι ισοσκελισμένοι και με το 3-pack και με το 6-pack και με το δημοσιονομικό σύμφωνο. Όλοι προσπαθούμε να οδηγηθούμε στους ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς και θα συμφωνήσουμε σε αυτό. Όμως από την άλλη, ε, και εδώ είναι η πρόκλησή μου αν θέλετε, χωρίς την οικονομική ανάπτυξη δεν μπορεί να υπάρξει δημοσιονομική εξυγίανση με την έννοια ότι μπαίνουμε σε ένα φαύλο κύκλο πράγματι. Αν δεν μπορούμε να καταλάβουμε ότι αν μπούμε σε μία βαθιά ύφεση τότε δυστυχώς δεν θα είναι ποτέ επαρκής οι περικοπές τις οποίες θα κάνουμε και θα πω στην κυρία Ποδήματα την οποία εκτιμώ ιδιαίτερα και την ακούω πάντα στις σκέψεις τις οποίες εκφράζει πέρα από τις ε, ιδεολογικές διαφορές υπάρχει ένα επίπεδο το οποίο ε, θα έλεγα με κάνει να ακούω με προσοχή αυτά τα οποία λέγει. Θα ήθελα λοιπόν να μου επιτρέψετε να είμαι εδώ λίγο προκλητικός. Δεν θα πρέπει εμείς να πιστεύουμε σε χώρες όπως την Ισπανία, την Ιταλία και την Ελλάδα ότι μπορούμε να πιέζουμε μόνο τις επιχειρήσεις ή και την ίδια τη Γαλλία που έχει μια πολύ ισχυρή φορολογική πίεση προς τις επιχειρήσεις. Μπορεί κανείς με ισχυρές τέτοιες πιέσεις ή στις οικογένειες, στις επιχειρήσεις, σε όλους τους οικονομικούς εταίρους να προχωρήσουμε. Ξέρουμε ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις χώρες, αλλά το σύστημα αυτό το οποίο επηρεάζει τις επιχειρήσεις, επηρεάζει τις οικογένειες, οδηγεί στην ύφεση ή οδηγεί στην ανάπτυξη. Μήπως θα ήταν πιο σωστό να περικόψουμε τη δημόσια δαπάνη, ακόμα και στις περιφέρειες, ακόμα και στις επαρχίες, ακόμα και στους δήμους, Υπάρχει θα έλεγα εδώ μια διάσταση η οποία πρέπει να διορθωθεί, πρέπει να αντιμετωπιστεί. Ο κύριος Γκίγκολτ σε αυτά είναι πολύ ευαίσθητος. Ε, η κατάσταση που επικρατεί σε ορισμένες περιφέρειες λόγω της φορολογικής και δημοσιονομικής αποκέντρωσης έχει δημιουργηθεί μια κατάσταση η οποία μας φοβίζει. Λοιπόν, ας καταλήξουμε ότι πρέπει να προχωρήσουμε σε περικοπές πρώτα στον δημόσιο τομέα γιατί συγκεκριμένα στο δημόσιο τομέα σοβούν καταστάσεις απαράδεκτες πολλές φορές. Είμαι λοιπόν έτοιμος να, να δω τις τροπολογίες σας, όλες τις έξυπνες προτάσεις οι οποίες θα προέλθουν από όλους τους συναδέλφους, λαμβάνοντας υπόψη ότι ε, προέρχονται ίσως από σχολές σκέψεις διαφορετικές από τη δική μου και ότι εγώ προέρχομαι από μια σχολή σκέψης η οποία μου λέει ότι για να φύγουμε από την κρίση θέλουμε την ανάπτυξη. Το θέμα είναι να βρούμε το σωστό δρόμο για την ανάπτυξη. Ευχαριστώ κύριε Παλώνε. Σας θυμίζω ότι η προθεσμία κατάθεσης είναι... 19 του μηνός. 6 Οκτωβρίου και 28 Οκτωβρίου θα γίνει συζήτηση των τροπολογιών αλλά και η ψηφοφορία στην Ολομέλεια των... Δεκέμβριο, αν θέλει ο Θεός. Έχουμε εξαντλήσει τα σημεία της ημερήσιας διάταξης για σήμερα. Αύριο θα έχουμε την ακρόαση για την Τραπεζική Ένωση, τα θέματα της ε, επίλυσης και της εποπτείας. Αύριο το πρωί στην 3 σε 50. Καλό βράδυ σε όλους και όλες.